Καθίστε συνάδελφοι. Δεν είμαστε αρκετοί. Υπάρχουν πολλοί απόντες δυστυχώς. Θα πρέπει όμως να σεβαστούμε λίγο το χρόνο για τον φιλοξενούμενό μας και για όλους που είναι από την αρχή εδώ. Με πάρα πολύ μεγάλη χαρά λοιπόν, αγαπητέ κύριε Υπουργέ, σας καλωσορίζω για δεύτερη φορά. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα η στιγμή, όχι μόνο γιατί θα εμβαθύνουμε από κοινού στα θέματα τα οποία θα συζητηθούν στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων, το οποίο έγινε στις 7 και 8 του μηνός, αλλά θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε σε ένα ενδιαφέροντα θα έλεγα διάλογο και να σχολιάσουμε τα αποτελέσματα της Σουηδικής Προεδρίας και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και να σας συγχαρώ για τις ιδιαίτερα στενές σχέσεις και σχέσεις συνεργασίας τις οποίες είχατε μαζί μας, ήσασταν πάντα πρωταγωνιστής της συνεργασίας αυτής. Την Δευτέρα και την Τρίτη αυτή της εβδομάδας το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων και Εξωτερικών Υποθέσεων συζήτησε κάποια από τα θέματα, θα αναφερθείτε σε κάποια από αυτά, όχι αναλυτικά σε όλα βέβαια, και η συζήτηση νομίζω θα εμβαθύνει τα θέματα αυτά. Υπάρχει το θέμα της ε, ολοκλήρωση στην Ευρωπαϊκή Ένωση των Δυτικών Βαλκανίων. Εκεί έχουν γίνει πολύ σημαντικές προσπάθειες για την κατάληξη σε συγκεκριμένα κριτήρια σχετικά με την Κροατία. Υπάρχουν επίσης και θετικά μηνύματα σχετικά με την τέως Ιουκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, λέει ο μιλητής που δεν οδήγησαν βέβαια σε μια συγκεκριμενοποίηση της ημερομηνία για την έναρξη των διαπραγματεύσεων. Υπήρξαν φυσικά και άλλα θέματα που αφορούν άλλες χώρες της περιοχής, ειδικά η δύσκολη περίπτωση της Βοσνίας Ευζεγοβίνης, η οποία βρίσκεται σε μια κατάσταση η οποία θα έλεγα δημιουργεί ορισμένες ανησυχίες, αν και υπάρχουν και κάποια θετικά στοιχεία στα οποία επίσης θα μπορούσαμε να σταθούμε. Υπάρχει επίσης και η ευαίσθητη θέση στην οποία κατέληξε το Συμβούλιο σχετικά με την Τουρκία και το βασικό χαρακτηριστικό κριτικής των σχέσεων της Τουρκίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση, η εξομάλυνση των σχέσεων της χώρας αυτής με την Κυπριακή Δημοκρατία. Υπάρχει επίσης και το θέμα το πολύ ευαίσθητο της ειρηνευτικής διαδικασίας στην Μέση Ανατολή. Το Συμβούλιο εξεφράστη πολύ συγκεκριμένα, θα έλεγα, σαφέστατα ευανάγνωστες οι θέσεις του Συμβουλίου, όχι μόνο υπάρχει ανάγκη να ξεκινήσει εκ νέου μια ειρηνευτική διαδικασία για τη δημιουργία δύο ανεξαρτήτων κρατών ικανών να ζήσουν και να ζήσουν μαζί μάλιστα το ένα δίπλα στο άλλο, με εγγυημένα σύνορα και με πλήρη διεθνή νομιμοποίηση. Αλλά καταλήξατε επίσης και σε μία θέση σαφέστατη, η οποία προκάλεσε πάρα πολλές αντιδράσεις από τα διάφορα εμπλεκόμενα μέρη, σχετικά με την πόλη των Ιεροσολύμων, η οποία θα πρέπει να είναι κατά το Συμβούλιο πρωτεύουσα δύο κρατών. Πώς θα προχωρήσει από εδώ και πέρα λοιπόν. Νομίζω ότι εδώ ίσως προκαταλαμβάνω κάποιες περίπλοκες ερωτήσεις των συναδέλφων που θα ακολουθήσουν, αλλά μετά από τις δηλώσεις και των Αμερικανών για την Ιερουσαλήμ πρωτεύουσα των δύο κρατών, πρόκειται για δηλώσεις οι οποίες δεν είναι οι τελικές, είναι προσωρινές, αλλά νομίζω ότι μπορούμε να προχωρήσουμε και προς τα εκεί. Έχουμε και την διαδικασία εκδημοκρατισμού του Ιράκ, οι εκλογές οι οποίες καθορίστηκαν για την 7η Μαρτίου του 10 και ο ρόλος της Ένωσης γύρω από την υπόθεση αυτή. Υπάρχει επίσης και το θέμα της εταιρικής σχέσης ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Λατινική Αμερική. Τίτλους σας έδωσα, λέει ο κ. Αλμπερτίνη, για να ορίσω λίγο το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα αναπτύξετε εσείς τα σημαντικά θέματά σας. Και που είναι ο βασικός στόχος λοιπόν της παρουσίας σας εδώ. Σας ευχαριστώ λοιπόν, φτάσατε ε, πραγματικά έγκαιρα. Η ακρίβεια αυτή χαρακτηρίζει θα έλεγα τον τρόπο με τον οποίο προεδρεύετε και σας δίνω τον λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πράγματι είναι μεγάλη χαρά να βρίσκομαι εδώ πέρα σήμερα. Πράγματι εκτίμησα κάθε ευκαιρία που είχα να συναντηθώ με τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του, Κοινοβουλίου είτε εδώ είτε στο Στρασβούργο, είτε σε ε, μεμονωμένες συζητήσεις. Ε, αυτό αποτέλεσε σημαντική συμβολή στη δουλειά της Προεδρίας μας. Επίσης μπορώ να σας πω ότι στο διάστημα που προείδρευσα στο Συμβούλιο προσπάθησα να, ε, ε, ε επιβάλλω ε, την ε, πειθαρχία των βορείων χωρών, αλλά κάτι τέτοιο δεν το κατάφερα. Φαίνεται να είναι η ασθένεια των Βρυξελών. Θα πρέπει να το δουλέψουμε αυτό τα επόμενα χρόνια. Ίσως η συνθήκη της Λισαβόνας να επιφέρει κάποια αλλαγή. Σύντομα να σας πω τι κάναμε κατά τη διάρκεια της Σουηδικής Προεδρίας. Τονίζοντας όμως ότι δεν έχει ε, ολοκληρωθεί η Σουηδική Προεδρία, θα ε, διατηρήσουμε την ε, πλήρη επιχειρησιακή ευθύνη για την ε, κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας μέχρι να χτυπήσουν οι καμπάνες την παραμονή το, της πρωτοχρονιάς. Ο κόσμος κινείται γρήγορα, μπορεί ακόμα να συμβούν πράγματα. Θυμάμαι την τελευταία φάση της γαλλικής προεδρίας όπου ξεκίνησε πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Δεν περιμένω κάτι τέτοιο, αλλά έπρεπε να συγκληθούν οι υπουργοί ε, το βράδυ πριν την παραμονή το, της ε, πρωτοχρονιάς. Ε, το είπα αυτό στους αδέρφους μου χθε το βράδυ. Δεν νομίζω ότι δεν τους άρεσε που το, το είπα, αλλά είναι γεγονός ότι μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. όταν κοιτούσα μπροστά τον Ιούλιο, βρισκόμασταν σε πολύ δύσκολη θέση και σε μια πολύ σημαντική στιγμή στην για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αντιμετωπίζαμε ε, οικονομική κρίση τέτοιου μεγέθους που βλέπει κανείς ε, μια φορά ε, στη ζωή του και αντιμετωπίζουμε και κρίση στο κλίμα από τέτοιες που βλέπει κανείς μια φορά αναχιλιετία. Δεν θα πω σε λεπτομέρειες σχετικά με τα οικονομικά και νομισματικά θέματα. Θα θυμάστε όμως ότι ανησυχούσαμε για τις επιπτώσεις τους στην ε, πολιτική ασφαλείας. Αυτή τη στιγμή πατάμε σε πιο σταθερό έδαφος ε, στις περισσότερες ε, χώρες που είχαν, για τις οποίες ανησυχούσαμε περισσότερο. Ε, χάρη στις ε, προσπάθειες ε, της Σουηδικής Προεδρίας πρέπει να πούμε, παρακολουθήσαμε στενά την κατάσταση, ήμασταν έτοιμοι να βοηθήσουμε και νομίζω ότι δημιουργήθηκε ένα κλίμα εμπιστοσύνης. Το κλίμα, πρόκληση, βρισκόμαστε στις τελευταίες μέρες ε, για την ε, προετοιμασία της ε, διάσκεψης υψηλού επίπεδου της Κοπενχάγης. Ήδη έχουν ξεκινήσει οι προετοιμασίες. Η διάσκεψη κορυφή στην Κοπενχάγη λοιπόν θα γίνει στο τέλος της επόμενης εβδομάδας. Εγώ θα βρεθώ εκεί από την αρχή της εβδομάδας για να συζητήσω τις μακροπρόθεσμες συνέπειες για την ασφάλεια. Θα συζητήσω συζητήσουμε το θέμα αυτό και απόψε στο γεύμα, καθώ και αύριο που θα συζητήσουμε τον ηγετικό ρόλο που έχει αναλάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση στον τομέα του κλίματο. Ε, γενικά, πάντω ε, έχουμε μια αισιοδοξία. Μπορεί να μην πετύχουμε όλα όσα ζητήσουμε, δεν λειτουργεί έτσι ο κόσμο, αλλά νομίζουμε ότι ε, θα πετύχουμε πρόοδο. Είμαστε συγκρατημένα αισιόδοξοι και η δουλειά που μας περιμένει τις επόμενες μέρες δεν θα πρέπει να, με κανένα τρόπο να υποτιμηθεί. Άλλα θέματα που συζητήσαμε τον Ιούλιο ε, ήταν μεταξύ άλλων η διεύρυνση και τον Ιούλιο τόνισα ότι η αξιοπιστία μας στον υπόλοιπο κόσμο βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην δυνατότητά μας ε, να προστατεύσουμε την ειρήνη και την ευημερία της ε, δικής μας ε, περιοχής. Αν δεν το πετύχουμε αυτό εδώ πέρα δεν θα έχουμε αξιοπιστία πουθενά ο υπόλοιπος κόσμος βλέπει την επιτυχία μας ε, στην πατρίδα μας ε, σαν ε, το αποφασιστικό τεστ για την επιτυχία μας και για την αξιοπιστία μας. Τον Ιούλιο θα θυμάστε ότι ανησυχούσα για την κατάσταση που αντιμετωπίζαμε. Είχαμε αρκετά εμπόδια στην διεύρυνση που όλα μαζί κινδύνευαν να να οδηγήσουν σε πολύπλοκες ε, καταστάσεις. Δεν θα έλεγα ότι λύσαμε όλα τα προβλήματα, δεν τα λύσαμε. Ε, υπάρχουν ακόμα κάποιες σημαντικές προκλήσεις ε, που παραμένουν και θα αναφερθώ, μπορώ να αναφερθώ σε αυτές, αλλά σίγουρα βρισκόμαστε σε καλύτερη θέση τώρα από ό,τι πριν από κάποιους μήνες. Η κροατική προσχώρηση προχωράει στην ε, τελευταία διάσκεψη για την ε, προσχώρηση που ε, είχαμε με τους Κροάτες. Κλείσαμε 8 κεφάλαια και ανοίξαμε άλλα 8. Έχουμε προχωρήσει λοιπόν πολύ σε σχέση με το ε, απόλυτο μπλοκάρισμα που αντιμετωπίζαμε στην αρχή της Σουηδικής Προεδρίας. Με το Μαυροβούνιο. Ε, έχουμε προχωρήσει, έχουμε στείλει την αίτηση της ε, Αλβανίας. Φαντάζομαι ότι κάποια στιγμή κατά τη διάρκεια της επόμενης ε, χρονιάς θα καταλήξει η αίτηση στο τραπέζι του Συμβουλίου και το Μαυροβούνιο χθες ή προχθές, ε, είπαμε τη σχετική αίτηση. Η Σερβία έχει συζητηθεί πολύ. θα σημειώσατε όμως ότι μπορέσαμε να άρουμε το μπλοκάρισμα στην εφαρμογή της ε, ε, συμφωνίας ε, και το αργότερο μέσα σε έξι μήνες θα ξεκινήσει η εφαρμογή του, της SAA. Όσον αφορά την Μακεδονία, λέει ο μιλητής, και το θέμα αυτό συζητήθηκε αρκετά προχθές τις προάλλες σημειώσαμε τη θέση του Συμβουλίου ε, στην ε, πολύ θετική ε, αξιολόγηση του, του, της Κομισιόν και είπαμε ότι θα επανέλθουμε στο θέμα αυτό τους επόμενους μήνες κατά τη διάρκεια της Ισπανικής Προεδρίας. Σημειώσαμε το πολύ θετικό κλίμα που υπάρχει στις διμερείς σχέσεις Σκοπίων και Αθηνών. Νομίζω ότι υπάρχει πιο θετικό κλίμα, αλλά να προσθέσω επίσης ότι εάν αυτό το πιο θετικό κλίμα δεν μετατραπεί σε συγκεκριμένες συμφωνίες μέσα στους επόμενους μήνες, φοβάμαι ότι θα χάσουμε αυτό το παράθυρο ευκαιρίας και θα βρεθούμε σε πιο δύσκολη θέση. Το λέω αυτό σε όλους σας. Και το λέω αυτό και σε αυτούς στους οποίους θα παραδώσω την σκητάλη την 1η Ιανουαρίου. Η Βοσνία είναι κάπως πιο προβληματική όπως όλοι γνωρίζουμε. Πολύ χρόνο δαπανίσαμε με τους ηγέτες της Βοσνίας. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλη χώρα με την οποία ε, πέρασα τόσο χρόνο ε, φέτος. Τέσσερις ολοήμερες συνεδριάσεις είχαμε τους ε, ηγέτες ε, της Βοσνίας για να πετύχουμε συμφωνία σε κάποια ελάχιστα πράγματα για να μπορέσουν να μπουν σε μια νέα φάση στην ε, διαδικασία προσχώρησης. Ε, ε, επειδή αναμένονται εξελίξεις του χρόνου στη Βοσνία, αυτό φαίνεται να είναι σημαντική πρόκληση. Σε στενή συνεργασία με τους Αμερικανούς φίλους μας έχουμε καταβάλει προσπάθειες. Ο Αμερικανός συνάδελφος ήταν εκεί τρεις φορές, εγώ, όπως και εγώ άλλωστε. Έχω πάει αρκετέ φορέ. Πάντω ε, η κατάσταση στα Δυτικά Βαλκάνια ε, που πριν από έξι μήνες ε, χαρακτηριζόταν από πλοκάρισμα τώρα πια χαρακτηρίζεται μάλλον περισσότερο από κάποιες εξελίξεις. Τουρκία. Για να παραμείνουμε στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Και εδώ προχωράμε, προοδεύουμε. Είχαμε πολύ καλή συζήτηση για την προσχώρηση της Τουρκίας και στο Κοινοβούλιο, στο Στρασβούργο την προηγούμενη εβδομάδα και στο Συμβούλιο Δευτέρα βράδυ Τρίτη. Συζήτηση που ήταν πολύ περισσότερο στρατηγικής φύσης από ό,τι συνήθως. Φυσικά μας ανησυχεί και το γεγονός ότι η Τουρκία δεν έχει εφαρμόσει το πρωτόκολλο της Άγκυρας. Ε, ελπίζουμε όμως ότι οι συνομιλίες για την Κύπρο θα προχωρήσουν με τέτοιο τρόπο ώστε να βρεθούμε σε νέα κατάσταση μέσα στους επόμενους μήνες σε αρκετούς ε, τομείς. 21 ε, Δεκεμβρίου ε, θα γίνει η διάσκεψη και περιμένουμε εκεί νέα σημάδια της προσχώρησης της Τουρκίας. υπεγράφει πρωτόκολλο με την Αρμενία τους περασμένους ε, μήνες και υπάρχει και η λεγόμενη δημοκρατική ε, πρωτοβουλία η οποία έχει να κάνει με τα δικαιώματα των Κούρδων ε, και υπάρχουν και κάποιες άλλες πρωτοβουλίες περιφερειακής πολιτικής και εξωτερικής πολιτικής που έχει αναλάβει η τουρκική προεδρία που δείχνουν την πρόοδο που σημειώνεται. Όσον αφορά την προσχώρηση, επιτρέψτε μου επίσης να σημειώσω την αίτηση προσχώρησης της Ισλανδίας την οποία υποβάλαμε στην Κομισιόν. Η Ισλανδία απάντησε στο ερωτηματολόγιο και περιμένουμε από την Κομισιόν να αναφέρει τα αποτελέσματα στο Συμβούλιο τους επόμενους ε, μήνες. Ε, στα συμπεράσματα του Συμβουλίου είπαμε ότι όταν γίνει αυτό το Συμβούλιο θα πρέπει να είναι έτοιμο να χειριστεί την αίτηση, δηλαδή να ανοίξει τις διαπραγματεύσεις για την προσχώρηση τον Ιούλιο. Το είπα και νομίζω ότι είναι σημαντικό να το επαναλάβω. Όλες αυτές οι προσχωρήσεις και οι εταιρικέ σχέσεις ε, ε, στην περιοχή μας ανοίγουν στρατηγικές προοπτικές. Οι περισσότερες συνδέονται με την ε, ε, νοτιοανατολική Ευρώπη, αλλά σαν Ευρωπαϊκή Ένωση ε, το να δραστηριοποιηθούμε στον ε, Υψηλό Βορρά και σε θέματα Αρκτικής έχει και αυτό μεγάλη στρατηγική σημασία. Στο Συμβούλιο τον, την Τρίτη Είχαμε έγγραφο ε, πολιτικής και στρατηγικής κατεύθυνσης για τις αρκτικές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και αυτό είναι ε, ένα νέο σημαντικό θέμα που έγινε τους τελευταίους μήνες. Είχαμε επιτυχίες και αποτυχίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είχαμε σχεδιάσει μια μεγάλη υπουργική διάσκεψη στην Κωνσταντινούπολη που δεν πραγματοποιήθηκε. Αυτό ήταν μια αποτυχία. Αυτό οφείλεται στο γνωστό γεγονός ότι οι ε, Υπουργοί Εξωτερικών ε, δεν είναι διατεθειμένοι να ε, συνομιλήσουν με τον Υπουργό Εξωτερικών του του Ισραήλ. Δυστυχώς λοιπόν αναγκαστήκαμε να κυρώσουμε τη συνάντηση αυτή προς μεγάλη μας λύπη. Σημειώνω Ελπίζω να μπορέσει να σπάσει ε, αυτός ο ε, φραγμός σύντομα ε, όσον αφορά την Υπουργική Διάσκεψη της Μεσογείου. Πέντε υπουργοί είχαν αρνηθεί να συμμετάσχουν. Πρόκειται λοιπόν για υπουργικό επίπεδο, για πρόβλημα σε υπουργικό επίπεδο. Η Τσεχική Προεδρία στην Πράγα ξεκίνησε Επίσης μια πρωτοβουλία που είχε να κάνει με το Φόρουμ της Κοινωνία των Πολιτών, ε, πολύ καλή συνάντηση πριν, κάποιους, πριν κάποιες εβδομάδες στις Βρυξέλλες και την Τρίτη είχαμε την ε, πρώτη υπουργική διάσκεψη της ε, Ανατολικής Εταιρικής ε, Σχέσης. Ήταν πολύ καλή η συνάντηση αυτή. Ξέρετε ότι πολλές από τις συναντήσεις που έχουμε γίνονται ως εξή. Έρχονται οι υπουργοί, βλέπουν τα έγγραφα που έχουν ετοιμάσει οι υπάλληλοι και μετά φεύγουν. Στη συγκεκριμένη περίπτωση όμως είχαμε μια ασυνήθιστα επικοδομητική συνάντηση με έξι υπουργούς εξωτερικών και εκπροσώπους του του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλους, οι οποίοι παρουσίασαν ιδέες και επέδειξαν ε, ένα επίπεδο αφοσίωσης στην ανάπτυξη ε, της ε, ανατολικής εταιρικής σχέσης που ξεπέρασε τις προσδοκίες πολλών. Δημιουργήσαμε διάφορες θεματικές πλατφόρμες, πρωτοβουλίες και έχουμε νέα θέματα και νέες πρωτοβουλίε μετά την συνάντηση της Τρίτης, ε, τις οποίες θα πρέπει να αναπτύξουμε περαιτέρω. Επιτρέψτε μου επίσης να αναφέρω ότι η πρόταση για την εντολή για τις συμφωνίες σύνδεσης του Νότιου Καυκάσου επίσης έχουν υποβληθεί. Ε, αναφέρθηκα σε αυτές τον ε, Ιούλιο. Ε, με τη Γεωργία ε, έχουμε ε, ετοιμάσει την Συμφωνία διευκόλυσης των Θεωρήσεων με τη χώρα αυτή που έχει ιδιαίτερη σημασία και πιστεύω ότι θα είναι δυνατόν να ανοίξουμε τις διαπραγματεύσεις με τη Γεωργία τους επόμενους μήνες. Θα ξεκινήσουμε τις διαπραγματεύσεις με τη Μολδαβία ε, πάνω σε μια συμφωνία σύνδεσης ε, μετά τις εκλογές και τις ε, πολιτικές αλλαγές που έγιναν εκεί ήταν σημαντικό με το μεγάλο άνοιγμα προς την Ευρώπη που αντιπροσώπευαν αυτές ήταν πολύ σημαντικό να στείλουμε ένα σημαντικό μήνυμα. Βρέθηκα εγώ εκεί και άλλοι και γι' αυτό ε, συμφωνήσαμε να ξεκινήσουμε τι διαπραγματεύσει αυτές. Θα ξεκινήσουν στις 21 Δεκεμβρίου και ως μέρος αυτών θα ξεκινήσει και διάλογος για τα θέματα ε, θεωρήσεων. Και η Ουκρανία είναι σημαντική. Είχαμε μια διάσκεψη κορυφή εκεί τι προάλλε θα, 17 Ιανουαρίου θα γίνει ο πρώτος γύρος των προεδρικών εκλογών ε, και ο δεύτερος γύρος θα γίνει στις 7 Φεβρουαρίου. Είχαμε πολύ καλή διάσκεψη κορυφής μαζί τους ε, με τον πρόεδρο Ιουσένκο, με την ε, πρωθυπουργό Τιμοσένκο και με τον κύριο Γιανκόβιτς που είναι ηγέτης της αντιπολίτευσης. Σε σημαντική ε, εκεί θα είναι η συνάντηση των Υπουργών Υγείας που θα πραγματοποιηθεί ε, στις 13 Δεκεμβρίου. Και ελπίζω πραγματικά ότι θα μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε τη συμφωνία ε, για την προσχώρηση της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ενέργειας. Αυτό νομίζω θα έχει πολύ μεγάλη σημασία. Δεν θα μπω σε πολλές λεπτομέρειες ε, σχετικά με, την, ε, με τις σχέσεις μεταξύ ημών και Λευκορωσίας. Απλά θα... Θα πρέπει να πω ότι είχαμε αρκετό κρασί αλλά και αρκετό νερό για να ε, αραιώσουμε το κρασί. Είναι κάτι στο οποίο θα πρέπει να εργαστούμε περισσότερο. Οι στρατηγικοί διάλογοι με διάφορους παγκόσμιου παράγοντες είναι επίσημα σημαντικό θέμα, να αναφερθώ σε κάποιου από αυτούς. Ε, σημαντική είναι η σχέση με τις Ηνωμένε Πολιτείε ε, και νομίζω ε, ότι έχουμε εξαιρετικές σχέσεις με τις Ηνωμένε Πολιτείε, με την κυβέρνηση Ομπάμα. Είχαμε τη διάσκεψη κορυφή στις 3 Νοεμβρίου. Τυπικά, αλλά ουσιαστικά πρόκειτο για τρίμερη συνάντηση έντονων διαλόγων σε πολλά επίπεδα και, σε, και για πολλά θέματα. Με άλλους εταίρους, ε, με τις ε, δυνάμεις που τώρα αναδύονται ε, στον κόσμο. Είχαμε μια διάσκεψη κορυφής στην Νότια Αφρική στις 11 Σεπτεμβρίου. Είχαμε συνάντηση με τη Βραζιλία στις 6 Οκτωβρίου, με την Ινδία στις 6 Νοεμβρίου, με τη Ρωσία στις 11 Νοεμβρίου, Κίνα 13 Νοεμβρίου και όπως σας είπα είχαμε και τη συνάντηση με την Ουκρανία. Ε, σε όλες αυτές τις συναντήσεις επικεντρωθήκαμε στην ε, αλλαγή του κλίματος και στις προετοιμασίες για την Κοπεχάγη. Ήμασταν ε, η επικεφαλής ε, δύναμη στην παγκόσμια κλιματική διπλωματία. Δεν θα πετύχουμε όλα όσα θέλουμε στην Κοπεχάγη, αλλά είναι σίγουρο ότι οι προσπάθειες της Ευρώπης έχουν προωθήσει την ε, κλιματική ατζέντα με τρόπο που δεν θα είχε συμβεί εάν ε, δεν ε, είχαμε δραστηριοποιηθεί. Μακροπρόθεσμα είναι σημαντικό να δημιουργήσουμε στρατηγικές εταιρικέ σχέσεις με τις αναδυόμενες δυνάμεις. Πολύ καλή συνάντηση με την Βραζιλία, με την Ινδία, πολλά υποσχόμενη συνάντηση με την Κίνα και είχα την χαρά να μπορώ να πάω στην Τζακάρτα και να υπογράψω την Συμφωνία εταιρική σχέση με την Ινδονησία χώρα με πληθυσμό 1 ε, ε, τέταρτο του δισεκατομμυρίου και ε, με πολλές δυνατότητες. Επίσης, με την Νότια Κορέα που είναι επίσης χώρα μεγάλης ε, σημασίας ε, είχαμε συνομιλίες. Ο ρόλος ε, της Ευρώπης στις διάφορες περιφέρειες όπου υπάρχουν κρίσεις από την Παλαιστίνη μέχρι το Πούντζαπ. Έχουμε επικεντρωθεί σε μεγάλο βαθμό στο Αφγανιστάν όταν συναντηθήκαμε τον Ιούλιο. Ετοιμαζόμασταν για τις προεδρικές εκλογές της 20 Αυγούστου. Ξέραμε ότι πρόκειτο να είναι πολύπλοκο το ζήτημα αυτό και νομίζω και υποψιαζόμουν ότι θα τα ταπανίσω πολύ χρόνο στο θέμα του Αφγανιστάν, αλλά ε, και πάλι υποτίμησα την ε, σημασία. Τελικά πρέπει να ταπανίσω ακόμα περισσότερο χρόνο στο θέμα του Αφγανιστάν, ε, στα θέματα μετά τις εκλογές, την ανεξάρτητη εκλογική επιτροπή, τους Ευρωπαίους παρατηρητές και θα ήθελα να ευχαριστήσω τον ε, συνάδελφο που ανέλαβε την ε, αποστολή στο Αφγανιστάν ε, μέχρι την ανάλυση των καθηκόντων του κυρίου Καρζάη και ως μέρος της διαδικασίας αυτής περάσαμε πολύ χρόνο αναπτύσσοντας ένα ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Αφγανιστάν και το Πακιστάν. Νομίζω ότι τώρα πια θεωρείται δεδομένο από όλους και από τους στρατιωτικούς ότι το πρόβλημα του Αφγανιστάν δεν είναι κυρίω, δεν είναι καν στρατιωτικό θέμα. Θα πετύχουμε στο Αφγανιστάν μόνο αν έχουμε πολιτική και οικονομική ε, συμμετοχή εκεί, τουλάχιστον όσο σημαντική ήταν η στρατιωτική μας προσπάθεια. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό να συμπεριλάβουμε τα πολιτικά και οικονομικά στοιχεία. Και είναι σημαντικό να το θυμόμαστε αυτό και στις ε, συνομιλίες που έχουμε και με τις Ηνωμένε Πολιτείες ε, και με άλλους. Συνεχίζουμε τις συζητήσεις για το πώς θα οργανώσουμε το συντονισμό των ε, πολιτικών και των πολιτικών προσπαθειών στο Αφγανιστάν. και θέλουμε έναν εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Καμπούλ ε, ώστε να μιλάμε με μία φωνή, διότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μία πολυφωνία, καλές φωνές δεν λέω, αλλά το να τραγουδάμε όλοι ταυτόχρονα μπορεί να μην είναι πολύ καλό. Θέλουμε λοιπόν έναν σολίστα. Αυτό θα γίνει αργότερα. Όσον αφορά τη Μέση Ανατολή, κύριε Πρόεδρε. Και αυτό εξακολουθεί να είναι ανησυχία της Προεδρίας. Μπορούμε να μοιράσουμε ε, την ε, κατάσταση σε δύο φάσεις. Η πρώτη φάση κάλυψε τους πρώτους μήνες της ε, Σουηδικής Προεδρίας και νομίζω ότι θα μπορούσε να πει κανείς ότι στηρίξαμε τις προσπάθειες του Γερουσιαστή Μίτσελ και του Προέδρου Ομπάμα. Με τη νέα Αμερικανική κυβέρνηση μας άρεσε η προσέγγιση της νέας κυβέρνησης Ομπάμα. Δεν ε, βλέπαμε το λόγο να κάνουμε κάτι δικό μας. Στηρίξαμε τους Αμερικάνους, ε, προσφέραμε την υποστήριξή μας. Η δεύτερη φάση όμως ήταν κάπως πιο διαφορετική, διότι είχαμε ανησυχίες σχετικά με την ε, έλλειψη προόδου και με το μπλοκάρισμα που υπήρχε και νιώσαμε ότι υπάρχει ανάγκη συζητήσεων σε επίπεδο Υπουργών Εξωτερικών για να ακουστεί πιο δυνατά η φωνή της Ευρώπης και αυτό ε, έγινε με το Συμβούλιο για τη Μεσή Ανατολή. Την Τρίτη είχαμε θίξαμε κάποια θέματα και ε, αυτά θα αποτελέσουν τη βάση της δράσης ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σίγουρα η συζήτηση που έγινε για τα θέματα αυτά στην περιοχή έχει δείξει ότι ακούγεται η φωνή της Ευρώπης, μετράει η φωνή της Ευρώπης σε τέτοιο βαθμό που πολλοί ε, ε μάλλον ένιωσαν θετική έκπληξη. Θα προωθήσουμε λοιπόν τα θέματα αυτά και νομίζω ότι αύριο θα έχουμε τη συνάντηση της Τρόικας εδώ στις Βρυξέλλες ε, με, τις, ε, με την Παλαιστινιακή Αρχή για να συζητήσουμε τα θέματα αυτά. Προσπαθήσαμε να βρούμε ημερομηνία για συνάντηση Τρόικας με το Ισραήλ, δεν μας έχουν απαντήσει όμως ακόμα. Κάποια στιγμή θα πραγματοποιηθεί και αυτό. Ε, μέχρι τώρα πάντως δεν ήταν δυνατό κάτι τέτοιο. Ένα άλλο θέμα που μας πήρε πολύ χρόνο είναι το Ιράν. Ήμασταν ξεκάθαροι σχετικά με την έκφραση των ανησυχιών μας για τα ανθρώπινα δικαιώματα στο Ιράν. Είδαμε μια περαιτέρω χειροτέρευση τις τελευταίες ημέρες. Μετά από αυτά τα οποία συνέβησαν κατά τη διάρκεια των προεδρικών εκλογών, εκφράσαμε την λύπη μας για τις συνέπειες οι οποίες προκλήθηκαν. Είχαμε κάποιες επαφές και κυρίως το θέμα φυσικά των πυρηνικών όπλων, στα πλαίσια της διτής αντιμετώπισης την οποία ακολουθεί το Συμβούλιο μας οδήγησε στο να υιοθετήσουμε μια δήλωση η οποία είχε προπαρασκευαστεί από το Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών την Τρίτη. Έχουμε και την κατάσταση στην Ονδούρα. Ο κόσμος είναι πολύ μεγάλος όπως βλέπετε και εκεί έχουμε πολλές ανησυχίες. Να ευχαριστήσω εδώ την Ισπανική κυβέρνηση που είναι τμήμα φυσικά και της Τρόικα για ό,τι έχουν κάνει μέχρι τώρα εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Προεδρίας. Την Τρίτη υιοθετήσαμε την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για το κέρας της Αφρικής. Θα καθοδηγήσει τους επόμενους μήνες και τα επόμενα χρόνια την παρουσία μας εκεί, την πολιτική μας εκεί. Υπάρχουν και άλλα που έχω ξεχάσει προφανώς. Να αναφέρω ε, μία βασική ανησυχία την οποία είχαμε κατά τη διάρκεια της Σουηδικής Προεδρίας είναι το θέμα της διαδικασίας που οδήγησε τη συνθήκη της Λισαβόνας στην αποδοχή της από όλους. Εξηγήσαμε τις θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και προς τους ψηφοφόρους της Δημοκρατίας της Ιρλανδίας. Χρειάστηκαν λεπτές πολιτικές κινήσεις και σε άλλες χώρες ή σε άλλη χώρα, λέει ο μιλητής, έτσι ώστε να επικυρωθεί τελικά από όλους η συνθήκη. Υπήρξαν ευαίσθητες κινήσεις και σε άλλα θέματα, οι οποίες συνεχίζονται. Φυσικά τώρα έχει τεθεί σε ισχύ η συνθήκη της Λισαβόνας από την 1 του ε, μηνός Δεκεμβρίου. Βρισκόμαστε σε μια εντελώς μεταβατική φάση για τα συμβούλια, αν και είναι μια συμμετρικά θα έλεγα ε, εξελισσόμενη φάση. Ξεχωρίσαμε την Δευτέρα και την Τρίτη το γενικών υποθέσεων από τη μία, των εξωτερικών υποθέσεων από την άλλη. Το ένα συμβούλιο προεδρεύεται πάντα από την προεδρεύουσα κάθε φορά χώρα και θα παραδώσουμε τις εργασίες, αν θέλετε, ε, του άλλου συμβουλίου στην μονιμότερη προεδρία του συμβουλίου. Καλωσόρισα την Κάθριν Άστον Συζητήσαμε ήδη μαζί της τα θέματα της ε, διεύρυνσης γιατί άπτονται φυσικά ε, των θεμάτων των εξωτερικών υποθέσεων και τα συζητήσαμε μαζί της αυτά και τη Δευτέρα και την Τρίτη για να διευκολύνουμε αυτήν την μετάβαση στην οποία αναφέρθηκα. Θα δοθεί ιδιαίτερη σημασία τους επόμενους μήνες στην υπηρεσία εξωτερικής δράσης. Υπάρχουν αρκετά θέματα εδώ το Συμβούλιο τις τελευταίες ημέρες του μηνός Οκτωβρίου ενέκρινε την πρόταση την οποία είχε καταθέσει η Προεδρία μετά από διαπραγματεύσεις εντατικές με όλες τις χώρες για τις κατευθυντήριες γραμμές για την ίδρυση ε, της Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό θα γίνει αντικείμενο φυσικά περαιτέρω διαλόγου και με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τις κυβερνήσεις στα πλαίσια των προσπαθειών να λειτουργήσει πλήρως στη συνθήκη της Λισαβόνας. Αυτά είναι κάποια από τα θέματα, Πρόεδρε, με τα οποία ασχοληθήκαμε. Σίγουρα έχω ξεχάσει κι άλλα. Να υπογραμμίσω όμως αυτό το οποίο ξεκίνησα λέγοντας, Το να είναι κανείς υπεύθυνο για τις εξωτερικές υποθέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης σημαίνει ότι πρέπει να είναι πάντα σε επιφυλακή κάθε στιγμή της μέρας και της νύχτας γιατί ο κόσμος κινείται και ο κόσμος ε, ίσως να είναι πιο απαιτητικός, πιο προκλητικός αν θέλετε και η κατάσταση της, στη διεθνή σκηνή να είναι και λίγο πιο επικίνδυνη από ό,τι ήταν πριν μερικά χρόνια. Εν πάση περιπτώσει τα πράγματα εξελίχθηκαν όπως σας είπα και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε έτσι ώστε ε, τους επόμενους μήνες να περάσουν τα θέματα της αρμοδιότητάς μου, όσα από αυτά περάσουν, στην Κάθριν Άστον με τον πιο σταδιακό και ήρεμο τρόπο μια πολύ θα έλεγα λία μετάβαση, ήρεμη μετάβαση στις νέες δομές τους επόμενους μήνες. Αυτός είναι ο άμεσος στόχος μας. Ευχαριστώ Υπουργέ, γιατί πράγματι είχατε ένα συγκεκριμένο χρόνο στη διάθεσή μας λόγω των εργασιών μας, καταφέρατε όμως να προχωρήσετε σε βάθος στην ανακοίνωσή σας, όπως πάντα. Ας περάσουμε τώρα στις ερωτήσεις. Θα ήθελα εδώ, όπως πάντα, να πω ότι οι εργασίες μας προβλέπουν τον περιορισμό των παρεμβάσεών σας. Να σεβαστείτε παρακαλώ 1,5 λεπτό. Σεβερίν έχει το λόγο, 1,5 λεπτό. Κύριε Υπουργέ, ξέρω από την εμπειρία μου ότι οι Υπουργοί είναι πάρα πολύ ε, βαρετοί, είναι πάρα πολύ ε, αμφιλεγόμενα αυτά που λένε. Δεν είσαστε καθόλου βαρετός και σας ευχαριστώ για αυτό. Παρακολούθησα την ε, ε, απόδοσή σας κατά το Σουηδική Προεδρία και είμαι ευτυχής που διαπιστώνω ότι στις περισσότερες περιπτώσεις είχαμε την ίδια άποψη. Θα ήθελα μόνο να πω το εξής. Ελπίζω και μετά το πέρας της Σουηδικής Προεδρίας η χώρα σας και εσείς ο ίδιος θα διατηρήσετε και η Ευρώπη θα διατηρήσετε τον ενδιαφέρον σας προκειμένου να συνεχιστεί αυτή η όθηση στην ευρωπαϊκή διαδικασία. Τώρα, για πιο συγκεκριμένα θέματα. Όντως, ήταν πολύ σημαντικό το γεγονός ότι το Συμβούλιο εξήγαγε συμπεράσματα για την Μέση Ανατολή. Πάντα ζητούσαμε ε, να μιλάει με μία φωνή η Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό συνέβη επιτέλους. Ωστόσο, το, η ερώτησή μου είναι η εξής. Επειδή Λίγα προβλήματα, λίγα βασικά προβλήματα ουσιαστικά αναφέρθηκαν στα συμπεράσματα. Το θέματα των επικισμών και το θέματα της ασφάλειας δεν έλαβαν την αντιστοιχή προσοχή. Τι μπορείτε να πείτε για αυτά. Και μία ερώτηση για το Ιράν. Η Σουηδική Προεδρία τι μήνυμα θα αποστείλει για τις επόμενες προεδρίες ή την επόμενη προεδρία ή και για τον μόνιμο πρόεδρο ποια θα είναι το κληροδότημά σας, αν θέλετε. Για μια πιο, αν θέλετε, άκαμπτη και πιο συνεκτική πολιτική για το Ιράν. Ευχαριστώ, κύριε Σίβερεν. Ε, Ένα μισή λεπτό επόμενος ο μιλητής, ο κύριος Βάγκελ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μιλήσαμε για δύο θέματα. Θα ήθελα να μιλήσω για δύο θέματα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Μπίλτ καταρχάς για το δεύτερο τμήμα της εισαγωγής σας για το αμφιλεγόμενο αν θέλετε της ε, παρουσίασής σας. Νομίζω ότι καταφέρατε να παρουσιάσετε κάποια θέματα τα οποία προηγουμένως δεν είχαν παρουσιαστεί και χάρηκα που αναφερθήκατε στο θέμα της Ιερουσαλήμ και που ξεκινήσατε συζητήσεις οι οποίες ε, τελικά αποτέλεσαν ένα βήμα προς τα εμπρός. Ωστόσο, δεν ε, βλέπουμε να προδιαγράφεται μια συγκεκριμένη λύση ακόμα. Λοιπόν, ρωτώ, πώς μπορούμε να πείσουμε το Ισραήλ για το ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι αρνητικά διακείμενη απέναντι του, αλλά για, επίσης ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και η συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να έχει και ωφέλη για το Ισραήλ. Γιατί ήταν πολύ αρνητική έναντι των ε, πρωτοβουλειών μας ως τώρα και το Ισραήλ συχνά διακυβεύει τα πάντα στις σχέσεις μας. Και δεύτερη ερώτηση αναφορικά με τη Βοσνία Ζεγοβίνη. Φαίνεται ότι πλέον έχει έρθει το πλήρωμα του χρόνου να δημιουργηθεί μια νέα ομάδα επαφή στη Βοσνία Ζεγοβίνη, η οποία θα συνδράμει στην εξέβρεση μιας λύσεως από το διέξοδο αυτό σε ό,τι αφορά τις δραματικέ υποθέσεις. Και η δική σας εμπειρία εκεί ήταν αρκετά επίπονη, από όσο ξέρω. Ναι, λυπάμαι. Θα σας διακόψω, γιατί έχετε θέσει ερωτήσει και θα πρέπει να σεβαστούμε και τους άλλους συναδέλφου που έχουν να θέσουν ερωτήσεις. Ευχαριστώ, επόμενος ομιλητή. Ευχαριστώ και ευχαριστώ κύριο Στάραντ. Ε, ευχαριστώ Υπουργέ για την παρουσίασή σας αυτή. Ωστόσο, επειδή έχει και το Κοινοβούλιο τα καθήκοντά του, εγώ ως πράσινος θα ήθελα να εκφράσω κάποιες ανησυχίες υπό τη μορφή των ερωτήσεων. Να εξή ερωτήσεω. Γιατί αναβάλουμε και πάλι την έναρξη των διαπραγματεύσεων με τη Μακεδονία, λέει ο μιλητή. Και επίση, να σημειώσουμε ότι λέω Μακεδονία. Δεν χρησιμοποιώ το περιττό αυτό αρκτικό λέξο που χρησιμοποιείτε. Κατά δεύτερον, για την Κροατία. Τι πιστεύετε ότι πρέπει να κάνει ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση αν δεν συνεργαστεί με το δικαστήριο ε, η χώρα αυτή. Και κατά τρίτον, θεωρούμε ότι είναι καλό το γεγονός ότι ε, ξεκλείδωσε την ενδιάμεση αυτή συμφωνία με τη Σερβία το Συμβούλιο. Αλλά τι θα γίνει με τους θεσμούς της χώρας αυτής. Και τέλος, η Επιτροπή θα ξεκινήσει την διαδικασία απελευθέρωσης των θεωρήσεων με την Πρίστινα. Ευχαριστώ, κύριε Τάραντ. Ενάμιση λεπτό, κύριε Σκόβαλτ. E, e, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, άκουσα με μεγάλο ενδιαφέρον την παρουσίασή σας και σέβομαι ιδιαίτερα την εργασία, το έργο σας, ιδιαίτερα το πρόσφατο έργο σας. Να σας συγχαρώ για όσα έχετε πετύχει ως τώρα. Έχω δύο συγκεκριμένε ερωτήσει να θέσω. Η πρώτη για την ανατολική συνεργασία. Πρόκειται για μια επιτυχία την οποία προσωπικά αναλάβατε. Το έργο σας ήταν πολύ θετικό. Δεν έχω χρόνο ουσιαστικά να επιχειρηματολογήσω. Αλλά θεωρώ ότι το έργο αυτό δεν πάει τόσο καλά όσο μας λέτε. Θα μπορούσατε να μας δώσετε μια μη διπλωματική και αν θέλετε και επικριτική ε, αξιολόγηση για το σχόλιο αυτό, για το έργο αυτό, το πρόγραμμα αυτό. Πιστεύω στο πρόγραμμα, αλλά θεωρώ ότι ήταν μάλλον τεχνητά ε, αισιόδοξη η εκτίμησή σας. Και άλλη μια ερώτηση. Θα ήθελα προσωπικά να σας ρωτήσω το εξή. Θα ήθελα να μου πείτε την προσωπική σας άποψη. Ναι και κλείνω πρόεδρε. Την προσωπική σας άποψη θα ήθελα να μας πείτε για τον πολιτικό ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Αφγανιστάν. Τι πιστεύετε για τις δραστηριότητες τις οποίες θα πρέπει να λάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Ο κ. Χατζηγεωργίου, 1,5 λεπτό. Ah, ε, είναι εδώ κύριε Χατζηγεωργή, έχετε το λόγο. È andato, non c'è. Allora, eh, l'onorevole per e Ο κύριος Κλάιες, ένα μισή λεπτό. Eh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, θα ήθελα να θέσω κάποια ερωτήματα για την Τουρκία την οποία όλος παραδόξως ε, τοποθετήσατε στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Είπατε ότι η Τουρκία σε ό,τι αφορά την Τελωνιακή Ένωση με την Ευρωπαϊκή ε, Ένωση δεν τηρεί τις υποχρεώσεις της. Σωστά. Και επίσης να προσθέσω ότι αρνείται να αναγνωρίσει όλα τα υφιστάμενα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχει deadline έχει οριστεί η καταλεκτική ημερομηνία για την Τουρκία για να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της και ποια είναι αυτή αν έχει όντως οριστεί. Μία άλλη ερώτηση. Το Συμβούλιο πώς αποθετείτε για τη νέα εξωτερική πολιτική της Τουρκίας που προσεγγίζει το Ιράν και τη Συρία και υιοθετεί όλο και πιο αντιδυτικές, αντιευρωπαϊκές ε, νοοτροπίες. Επίσης, ε, να αναφέρω τα συγχαρητήρια που έδωσε ο Ερντογάν στον Αχμαντινιτζάντ μετά την εκλογή του. Και επίσης να παραπέμψω στην δήλωση του Ερντογάν για το πρινικό πρόγραμμα του Ιράν που δήλωσε ότι τα δυτικά κράτη τα οποία προβάλλουν ενστάσεις για το γεγονός ότι το Ιράν ενδεχομένως έχει ενδεχομένως και σχεδόν σίγουρα ε, αναπτύσσει όπλα δεν είναι συγκεκριμένες και δεν είναι και ειλικρινές γιατί έχουν και τα δυτικά κράτη πυρηνικά όπλα. Όλα αυτά είναι τουλάχιστον ανησυχητικά. Πώς τοποθετείτε λοιπόν το Συμβούλιο ως προς τις ε, δηλώσεις αυτές και πώς θεωρεί το Συμβούλιο ότι θα συνεχίσουν αυτές οι εξελίξεις. Ευχαριστώ. Τάλερ για 1,5 λεπτό. Ε, θα ήθελα να σας συγχαρώ για τον πλήρη κατάλογο των δραστηριοτήτων σας τους προηγούμενους μήνες και των επιτευγμάτωσαν επίσης τους τελευταίους πάντα πέντε μήνες. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και γιατί κάνατε προσπάθειες για να ξεπεραστούν τα εμπόδια στις σχέσεις Κροατίας Σλοβενία. Σχετικά με την Μακεδονία, λέει ο μιλητής, κάνατε ό,τι μπορούσατε για να προωθήσετε την υπόθεση αυτή και έχω εδώ δύο ερωτήσεις. Η πρώτη, πέραν της Ελλάδας και της ε, Κύπρου υπήρχε κάποιος άλλος που να ήταν κατά της έναρξης των διαπραγματεύσεων με την χώρα αυτή που είναι υποψηφία, θυμίζω, εδώ και τέσσερα χρόνια. Και αν ναι, ήταν τα επιχειρήματά τους. Δεύτερον, Κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων τέθηκε το θέμα διασφάλισης της ειρήνης και της σταθερότητας στην περιοχή. Γνωρίζουμε ότι η Μακεδονία, λέει ο μιλητής, είναι ιδιαίτερα εύθραυστη και ευάλωτη. Και συμφωνώ μαζί σας ότι είναι δική μας ευθύνη και δική μας ευθύνη να δώσουμε τις απαιτούμενες εγγυήσει έτσι ώστε να διασφαλίσουμε την ειρήνη στην περιοχή. Λοιπόν, ευχαριστώ κύριε Τάλερ. Κλείνει ο πρώτος γύρος των ομιλιών, των παρεμβάσεων και θα δώσω το λόγο στον κύριο Μπίλντ πριν προχωρήσουμε στον δεύτερο γύρο. Ευχαριστώ πολύ ε, τους βουλευτές. Ε, δεν ξέρω αν θα μπορέσω να απαντήσω σε όλα, θα προσπαθήσω πάντως. Ε, κύριε Σεβερίν, καταρχήν σας ευχαριστώ που είπατε ότι δεν είμαι βαρετός. Αυτό σίγουρα είναι κάτι. Θα λυπόμουν πάρα πολύ αν θεωρούσατε ότι είμαι βαρετός. Προτιμώ να είμαι ε, αμφιλεγόμενο πρόσωπο. Και δεν χρειάζεται να το πω αυτό σε ένα κοινοβούλιο. Ε, όντας κάποιος αμφιλεγόμενος κινεί τα πράγματα συχνά και Σίγουρα θα προσπαθήσω μέχρι το τέλος της Προεδρίας να είμαι ακόμα λιγότερο βαρετός από ό,τι μέχρι τώρα. Ας ξεκινήσουμε από τη Μέση Ανατολή. Και ο κύριος Βάγγελ είχε σχετική ερώτηση που συνδεόταν κυρίως με τη Γερουσαλήμ. Νομίζω ότι εξήγησα τις διάφορες φάσεις που έχει περάσει η πολιτική μας για τη Μέση Ανατολή. Αυτό που δεν κατάφερα. Αυτό που δεν έκανα ήταν να ε, επικροτήσω τις προσπάθειες ε, του Ξαβιέ Σολάνα κατά το διάστημα αυτό. Ε, δουλεύει, δουλεύει εδώ και αρκετό καιρό. Είχαμε πολύ καλές επαφές με όλους τους βασικούς παράγοντες. Είναι αποφασιστική σημασία τώρα να γίνει η κίνηση προς την κατεύθυνση ε, άμεσων διαπραγματεύσεων. Αυτό ήταν ε, αρκετά πιο δύσκολο από ό,τι είχαν προβλέψει αρκετοί άνθρωποι. Ε, υπήρχε αρχική επιφύλαξη από τη μια μεριά, τώρα υπάρχει επιφύλαξη από την άλλη μεριά. Πάντως ελπίζω ειλικρινά οι πολλοί σημαντική δήλωση, διακήρυξη που υιοθετήσαμε την Τρίτη να οδηγήσει στο ξεκίνημα άμεσων ε, συνομιλιών. Ε, δεν περιμένω αυτό να γίνει αύριο, αλλά είμαι ε, βέβαιος ότι όταν γραφτεί η ιστορία, η διακήρυξη της Τρίτης θα θεωρηθεί σημαντικό τούβλο στην προσπάθεια οικοδόμησης των άμεσων συνομιλιών. Την Τρίτη είπα ότι οι συνομιλίες αυτές θα πραγματοποιηθούν σε περιορισμένο χρονικό διάστημα. Τα ε, θέματα είναι γνωστά, δεν θα συνεχιστούν οι συζητήσεις επάπειρων. Ε, όλοι μας γνωρίζουμε ποια είναι η μόνη πιθανή λύση. Πολύ, πολλές συζητήσεις έχουν γίνει για το θέμα της ε, ε Σίγουρα ε, ξέρουμε όλοι ότι οι δραστηριότητες αυτές είναι παράνομες. έχουν γίνει κάποιες θετικές κινήσεις από την Ισραηλινή πλευρά, αλλά για ένα προσωρινό μορατόριο, αλλά αυτό δεν είναι όλα όσα ζήτησε η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά σίγουρα είναι περισσότερα από όσα έχουν γίνει μέχρι τώρα. Είναι κάτι που έχουμε σημειώσει θετικά. Η Ιερουσαλήμ ήταν ε, ε, στο επίκεντρο των ε, συζητήσεων το τελευταίο διάστημα, διότι ανησυχούμε πολύ με τις εξελίξεις εκεί και Ακόμα στις συζητήσεις που ελπίζουμε ότι θα ξεκινήσουν, εμείς ε, θέλουμε ως σημείο κίνησης ε, τα σύνορα πριν το 1967 συμπεριλαμβανομένες της Ιερουσαλήμ. Αυτό όμως από μόνο του λύνει το θέμα ε, της επίκησης με την εξαίρεση της Ιερουσαλήμ. Κάποια στιγμή το θέμα της Ιερουσαλήμ ε, θα αποτελέσει πυρηνικό θέμα στις ε, συνομιλίες και γι' αυτό είναι σημαντικό από την αρχή να ξεκινήσουμε την ε, θέση μας. Και μπορεί να είμαστε πιο ξεκαθαροί από άλλους, δεν θα πρέπει όμως να φοβηθούμε να είμαστε σαφείς, θα πρέπει να πούμε ότι δεν βλέπουμε άλλη λύση από αυτήν της Ιερουσαλήμ ως πρωτεύουσα σε δύο κρατών. Υπάρχουν πολλά δύσκολα θέματα, υπάρχουν ε, τα θέματα ασφαλείας. Ε, δεν έχουμε εκφραστεί, δεν έχουμε πάρει θέση σε όλα τα επιμέρους θέματα αλλά έχουμε εργαστεί με τα λεγόμενα αποθέματα. Ακούγεται σαν να είμαστε πελάτες σε τράπεζα, αλλά όταν ξεκινήσουν οι συνομιλίες, τι θα μπορεί να φέρει η Ευρώπη στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Μας ενδιαφέρει η οικοδόμηση του Παλαιστινιακού κράτους ο Πρωθυπουργό Αλεμφαγιάτ κάνει εξαιρετική δουλειά και στον τομέα τη ασφαλεία και αυτό αναγνωρίζεται και από την κυβέρνηση του Ισραήλ. Στην δυτική όχθη έχει σημειωθεί μεγάλη πρόοδο. Και αυτό ήταν σημαντικό για την προώθηση των οικονομικών δραστηριοτήτων ε, και υπήρξε άρση των ε, περιορισμών των Ισραηλινών στην δυτική όχθη που έχει συμβάλει στις ε, εξελίξεις. Έχει διευκολυνθεί δηλαδή η βελτίωση της οικονομικής κατάστασης. Όλα τα θέματα αυτά θα πρέπει να συζητηθούν και ε, εμείς ετοιμάζουμε τα θέματα αυτά των λεγόμενων αποθεμάτων ε, που θα μπορέσουμε, με τα οποία θα μπορέσουμε να συμβάλλουμε στον τομέα της ασφάλειας ε, και σε άλλους τομείς. Ο κύριος ε, μίλησε για τους όρους των Ισραηλινών. Ένα πράγμα να πω εδώ, ένα μήνυμα προς το Ισραήλ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχει. Δεν είμαι βέβαιο ότι ο Ισραηλινός τύπος εκφράζει τις θέσεις της ε, κυβέρνηση του Ισραήλ. Ελπίζω όχι. Αλλά, εάν διαβάσει κανείς τον Ισραηλινό τύπο, θα πίστευε κανείς ότι δεν υπάρχει η Ευρωπαϊκή Ένωση πιστεύουν ότι η σχέση με την Ευρώπη θα πρέπει να βασίζεται στο διέρη και βασίλευε. Δηλαδή, θεωρούν κάποιους καλούς και κάποιους κακούς και προσπαθούν να αποφεληθούν από τη θέση αυτή. Την Τρίτη, ε, αποδείχθηκε όμως ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχει και όσον αφορά τη Μέση Ανατολή. Και πιστεύω ότι στη διάρκεια του χρόνου, όσο εμβαθύνουμε στην ε, εφαρμογή της Λισαβόνας θα δείξουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ισχύει και ε, υπάρχει και αποτελεί σημαντικό παράγοντα σε όλα τα σημαντικά θέματα. Το παιχνίδι αυτό που παίζεται εδώ και χρόνια από κάποιους ε, θα έχει όλο και λιγότερα κέρδη. Θα φέρνει όλο και λιγότερα κέρδη σε αυτούς. Ο κύριος Σέβεριν και κάποιο... Ε, ε, απάντησα στον κύριο Σέβεριν, ο κύριος Κλέης αναφέρθηκε στο πυρηνικό θέμα, αναφέρθηκε και η Τουρκία. Έχουμε... Ε, βρισκόμαστε σε δημόσια συνεδρίαση τώρα. Είναι λοιπόν κάπως περιορισμένες οι συμβουλές που μπορώ να δώσω. Πάντως το θέμα αυτό είναι πάρα πολύ, είναι ιδιαίτερα πολύπλοκο. Κατά τη διάρκεια τη χρονιά είχαμε μια θετική και μια αρνητική εξέλιξη. Η θετική είναι φυσικά η νέα πολιτική της κυβέρνηση Ομπάμα. Εμείς οι Ευρωπαίοι Προσπαθούμε επί χρόνια να συνομιλήσουμε με το Ιράν για τα πυρηνικά θέματα. Ε, αλλά όταν οι Αμερικανοί μπήκαν στο παιχνίδι, βρεθήκαμε σε μια κατάσταση όπου μπορεί να επιτευχθεί κάτι ενδεχομένως. Και αυτό είναι πολύ θετικό. Ε, αλλά η αρνητική εξέλιξη δεν αφορά μόνο τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ε, καταπίεση. Αυτό ούτως ή άλλως είναι σημαντικό θέμα από μόνο του. Αλλά Πολύ σημαντικοί παράγοντες ε, στο Ιράν δεν ενδιαφέρονται να ξεκινήσουν επικοδομητικές συζητήσεις με τον εξωκόσμο. Δηλαδή, τη στιγμή που μπήκαν οι Αμερικανοί στο παιχνίδι και ε, ε, άνοιξαν κάποιες ευκαιρίες, το Ιράν βρίσκεται εσωτερικά σε δύσκολη θέση που δυσκολεύει την κατάσταση. Είχαμε... Κάποιες σημαντικές εξελίξεις. Εγώ πάντως δεν θα έκλεινα την πόρτα τώρα, αν και ο χρόνος ε, τελειώνει, ο χρόνος περνάει, διότι έχουμε τον ε, αντιδραστήρα του, ε, της Τεχεράνης, Υπάρχουν ακόμα σημαντικοί παράγοντες στο Ιράν που είναι διατεθειμένοι να συνομιλήσουμε. Βέβαια δεν είμαι ειδικό σε όλα τα εσωτερικά θέματα της ηγεσία στο Ιράν. Αλλά φαίνεται ότι αυτός είναι ο ένας παράγοντας που δυσκολεύει την κατάσταση. Θα πρέπει λοιπόν να συνεχίσουμε τις προσπάθειες και αν υπάρξει λύση στο θέμα αυτό θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε και σε πολλά άλλα θέματα. Το Ιράν είναι σημαντική χώρα. Εάν δεν υπάρξει πρόοδος θα πρέπει να εξετάσουμε τη χρήση άλλων μέτρων και θα πρέπει να τα εξετάσουμε με ψυχραιμία και με αναλυτικό τρόπο. Θα πρέπει να εξετάσουμε αν τα μέτρα αυτά είναι εφαρμόσιμα, εάν είναι αποτελεσματικά και αν θα συμβάλλουμε στην επίτευξη των πολιτικών στόχων που έχουμε θέσει. Το θέμα του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν ε, θα είναι θέμα εξαιρετικής σημασίας στους επόμενους μήνες. Ε, έχω ε, και κάποιες άλλες σκέψεις που θα μπορούσα να μοιραστώ μαζί σας, αλλά δεν νομίζω ότι μπορώ να το κάνω αυτό σε μια, δημόσια, σε μια ανοιχτή συζήτηση. Για τη Βοσνία, κύριε Βάικλ, έχουμε μια ομάδα επαφών με τη Βοσνία, έχουμε το ε, Συμβούλιο ε, το οποίο δημιούργησα εγώ πριν 15 ε, χρόνια, εμένα θα πρέπει να κατηγορήσετε δηλαδή, έχουμε καταβάλει προσπάθειες. Και πιστεύω ότι είναι σημαντική δουλειά. Έχουμε συνομιλήσει με Τούρκους, με τη Ρωσία στις προσπάθειες αυτές. Τούτου λεχθέντος όμως, υπάρχουν και θα πρέπει να υπάρχουν όρια για το τι μπορούμε να πετύχουμε στο συγκεκριμένο πλαίσιο. Ευρωπαϊκή Ένωση, ε, Ηνωμένε Πολιτείε, Τουρκία, σε κανέναν μας δεν, δεν ανήκει η Βοσνία. Ακόμα και στις δικές μας χώρες διαφωνούν οι πολιτικοί μεταξύ τους. Τελικά όμως, στις περισσότερες από τις χώρες αυτές καταφέρουμε να συμφωνήσουμε πάνω σε κάποια βασικά θέματα. Και αυτή είναι η τέχνη του απαραίτητου συμβιβασμού που θα πρέπει να ε, μάθουν και οι Βόσνοι. Οι, οι διεθνείς προσπάθειες ε, στην ε, Βοσνία θα πρέπει να πραγματοποιηθούν με πολύ προσοχή, διότι αν δεν γίνει αυτό τότε δεν ε, θα πετύχουμε αυτό το πνεύμα συμβιβασμού. Διότι θα είναι πιο, πολύ πιο εύκολο για τους πολιτικούς να συνεργαστούν με εξωτερικές δυνάμεις παρά να συμφωνήσουν με άλλους πολιτικούς της δικής τους χώρας. Πάντως ε, Είδα να συμβαίνει αυτό που συνέβαινε και πριν 10 χρόνια. Ε, να συνομιλεί ο κόσμος πολύ περισσότερο με τους ξένους τελικά. Όμως το μέλλον της Βοσνίας θα αποφασιστεί από την δυνατότητα των πολιτικών ηγετών της ε, Βοσνίας να συνομιλήσουν μεταξύ τους. Η Βοσνία ξέρει τι πρέπει να κάνει, θα πρέπει να τροποποιήσει το Σύνταγμα, θα πρέπει να ε, συμμορφωθεί με το ε, Διεθνές Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ε, και έχουμε και τις 5 συν 2 προϋποθέσεις για να κλείσει το γραφείο εκεί του υψηλού εκπρόσωπου. Και επανειλημμένα κατά τη διάρκεια της χρονιάς αυτής ε, έχω επαναλάβει την ανησυχία μου απέναντι στους ε, πολιτικούς ηγέτες ε, της Βοσνίας να κοιτάξουν την περιφέρεια. το, η Σερβία δεν θα είναι κλειστή για πάντα, η Αλβανία προχωράει, το Μαυροβούνιο προοδεύει και το είδαμε αυτό και στο θέμα της, των θεωρήσεων. Όταν ήμασταν εκεί ο Σφάτσενμπερ και εγώ τον Απρίλιο νομίζω, εγώ τους είπα, οι άλλοι προχωράνε, εσείς μένετε πίσω. Και αυτοί είπαν ότι ε, τι έγινε. Στις 19 Δεκεμβρίου ε, θα διευκολυνθούν ε, οι θεωρήσεις ε, για τους πολίτες του Φύρομ του Μαυροβουνίου. Αυτό είναι τραγικό για τη Βοσνία και ε, οφείλεται στην ε, ανικανότητα των Βοσνίων ηγετών να καταλάβουν κάποια πολύ βασικά πράγματα και υπάρχει ο κίνδυνος να συμβεί αυτό σε πολύ σημαντικότερα θέματα. Ελπίζω λοιπόν στην προεκλογή τους εκστρατεία να επικεντρωθούν λιγότερο στο παρελθόν και να επικεντρωθούν περισσότερο στο μέλλον. Όπω σα είπα, θα υπάρχουν διεθνεί δυνάμει εκεί για να βοηθήσουν και για να βοηθήσουν. Αλλά το σημαντικό είναι να στείλουμε ακριβώ αυτό το μήνυμα σε αυτούς. Γιατί φυρώμαι. Θα περιοριστώ λέγοντας αυτά τα οποία σας είπα και στην αρχή της ομιλίας μου. Εμείς εκπροσωπούμε την Ευρωπαϊκή Ένωση και υπάρχουν πολύ συγκεκριμένα όρια για το τι μπορούμε να κάνουμε. Μίλησα όμως και με τον κύριο Παπανδρέου και με τον κύριο Γκρουεύσκη ε, για το πώς ε, θα εξελίσσονται τα πράγματα και σε διμερές επίπεδο και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ελπίζω να προχωρήσουν οι διμερείς επαφές. Υπάρχουν πάντως συζητήσεις αυτή την εποχή που έχουν μια τέτοια φύση που στο παρελθόν δεν την είχαν. Είπατε ότι είναι μια εύθραυστη χώρα η Φιρόμ και περιμένει πολύ καιρό και της αξίζει να δώσουμε ένα θετικό μήνυμα. Μπορούμε να στείλουμε αυτό το μήνυμα στα πλαίσια των περιορισμών βέβαια τα οποία έχουμε σαν Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή Προεδρία των 27 χωρών. Οι επόμενοι μήνες εδώ μπορεί να είναι όμως πολύ σημαντικοί και ο ρόλος που θα παίξει η Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει σημαντικός. για την Ανατολική Εταιρική Σχέση. Ε, κάποιοι είπαν ότι ήμουν ιδιαιτέρως ε, ε, αισιόδοξο, τεχνητά αισιόδοξο. Αλήθεια είναι αυτό, είμαι περισσότερο αισιόδοξο μετά από την τελευταία συνάντηση που είχαμε την Τρίτη. Οι έξι υπουργοί ήρθαν και δεν είπαν τα συνηθισμένα, αλλά όλοι παρουσίασαν πρωτοβουλίες για το πώς να προχωρήσουν τα πράγματα. Αυτή η εταιρική σχέση λοιπόν προς Ανατολάς περνάει σε μια νέα φάση. Όλοι νιώθουμε ότι εμπλεκόμεθα πλέον σε αυτή τη νέα φάση. Βέβαια είναι ε, πολύ νωρίς ακόμα. Δεν έχουμε ξοδέψει καθόλου χρήματα. Τα χρήματα θα είναι διαθέσιμα έτσι και αλλιώς από την 1η Ιανουαρίου στα πλαίσια αυτή της εταιρική σχέσης προς Ανατολάς. Βρισκόμαστε δηλαδή σε μια αρχική φάση. Και αφού αρχίσουμε να δαπανούμε φυσικά τα χρήματα αυτά θα τεθεί το θέμα. Είναι αρκετά τα χρήματα. Πολλοί πιστεύουν ότι χρειάζονται περισσότερα. Δεν θα διαφωνήσω με αυτό. Και ένα από τα πράγματα τα οποία προσπαθούμε να κάνουμε και θα το μεταφέρω το θέμα αυτό και στην Ισπανική Προεδρία βέβαια διότι δεν ε, ε, ξεπερνάει τη χρονική διάρκεια μίας προεδρίας είναι τα οικονομικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να είναι πιο δραστήρια στην προσπάθεια αυτή την οποία κάνουμε προς Ανατολάς. Και αναφέρομαι εδώ και στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και στην έβρεση γενικότερα περισσότερων πηγών για την χρηματοδότηση των προγραμμάτων στα πλαίσια αυτής της πολιτικής γειτονίας. Λοιπόν, είναι περίπλοκα τα θέματα αυτά, υπάρχουν πάρα πολλές λεπτομέρειες, αλλά αυτά είναι τα βασικά θέματα με τα οποία ασχοληθήκαμε. Το θέμα των θεωρήσεων, σαν παράδειγμα. Αυτό που θέλουν όλες αυτές οι χώρες είναι η ελευθερία διακίνησης των πολιτών τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει λοιπόν να έχουμε μια πιο συγκεκριμένη αντίληψη, μια πιο ενιοποιημένη αντίληψη για τα θέματα των θεωρήσεων για τους κατοίκους των χωρών της ανατολικής πλευράς. Ίσως αυτές οι συζητήσεις βέβαια να γίνονται στα πλαίσια του Συμβουλίου Υπουργών Εξωτερικών Υποθέσεων και να υπάρχει μια κάποια συμφωνία εκεί, αλλά να μην ξεχνάτε ότι στο συγκεκριμένο θέμα υπάρχει και το Συμβούλιο Υπουργών Εσωτερικών Υποθέσεων που ασχολείται με τα θέματα των θεωρήσεων. Για την Τουρκία. Προφανώ. η Τουρκία είναι Νότια Ανατολική Ευρώπη και η Κύπρος είναι Νότια Ανατολική Ευρώπη. Δεν ανήκουν σε άλλο κόσμο η Κύπρος και η Τουρκία, έτσι δεν είναι. Στην Ασία ανήκει η Κύπρος. Α, όχι. Ε, τι θέλετε να πείτε, ότι η Κύπρος ανήκει στην Ευρώπη και η Τουρκία ανήκει στην Ασία. Διαρωτώ Η Τουρκία ανήκει σε αυτό που ονομάζουμε Μικρά Ασία, λέει ο Φλαμανδός βουλευτής. Και η Κύπρος που είναι. Είναι στην Ευρώπη, λέει ο Μπίλτ. Εγώ νόμιζα ότι η Κύπρος είναι πιο ανατολικά από ένα μεγάλο κομμάτι της Τουρκίας. Θα πρέπει να ξαναδώ τους χάρτες μου πάντως, λέει ο κύριος Μπίλτ. Εν πάση περιπτώσει και η Κύπρος και η Τουρκία έχουν καθοριστεί σαν τμήμα της Ευρώπης από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα και από το Συμβούλιο της Ευρώπης ε, για πάντα. Όχι βέβαια για πάντα, αλλά από τότε που έχουν λειτουργήσει οι οργανισμοί αυτοί και θα χρησιμοποιήσω την ορολογία τους αυτή. Ε, για την τουρκική εξωτερική πολιτική σε ορισμένου τομεί. Είναι αλήθεια ότι είναι πολύ πιο δραστήρια η Τουρκία στον τομέα τη εξωτερική πολιτική από ό,τι στο παρελθόν έχει μια εξωτερική πολιτική με τη δική της ταυτότητα, όπως η σουηδική εξωτερική πολιτική, η βρετανική εξωτερική πολιτική, καθορίζονται από την ιστορία τους, από το παρελθόν τους, από τα συμφέροντά τους. Και η Τουρκία προσπαθεί συστηματικά να μην έχει προβλήματα με τους ε, γείτονές της προς Ανατολάς, γιατί όχι. Κάθε χώρα έχει, θα έλεγα κάθε συμφέρον, να περιβάλλεται από ειρηνικές καταστάσεις Μερικές φορές κάποιοι γείτονες είναι ευχάριστοι, κάποιοι άλλοι είναι λιγότερο ευχάριστοι, αλλά γίνεται μια προσπάθεια να υπάρχουν σχέσεις με χώρες οι οποίες δεν παρουσιάζουν προβλήματα. Έχουν προχωρήσει στην εξομάλυνση των σχέσεων με τη Συρία οι Τούρκοι. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε και εμείς στις σχέσεις μας με τη Συρία. Έχουν πάρει πολύ ε, θαραλέα βήματα οι Τούρκοι απέναντι στην Τουρκία, στην Αρμενία, συγγνώμη. Ξέρετε, ο, πόνος που χωρίζει τις χώρες αυτές εδώ και πραγματικά πολύ καιρό και γι' αυτό χαιρετίζω το θάρρος των πολιτικών ηγεσιών της Τουρκίας και της Αρμενίας. Θα πρέπει βέβαια οι θέσεις αυτές να επικυρωθούν κοινοβουλευτικά και στις δύο χώρες και αυτό δεν θα είναι εύκολη στιγμή και για τις δύο χώρες και συνδέονται με πολλά άλλα θέματα. Έχουν επίσης συμφέροντα για καλές σχέσεις με το Ιράν. Αυτό συνδέεται επίσης και με, την κατάσταση στο Ιράκ. Θα είμαι ειλικρινής εδώ μαζί σας. Αν η Τουρκία και το Ιράν πρόκειται να έλθουν σε αντιπαράθεση σχετικά με τα θέματα του Βορείου Ιράκ, αυτό είναι κάτι που δεν θα επιτρέψει ποτέ να υπάρξει ειρήνη στη Μεσοποταμία. Η Τουρκία έχει προχωρήσει στην εξομάλυση των σχέσεων και με το Ιράκ και με την περιφερειακή κυβέρνηση του Αρμπίλ. Κανένας δεν πίστευε ότι κάτι τέτοιο θα ήταν εφικτό στο παρελθόν. Για το Ιράν τώρα και τα πυρηνικά όπλα δεν είναι καθόλου τυχαίο που ο κύριος Ερτοάν είχε πάει και συζητούσε αυτά τα θέματα στις αρχές της εβδομάδας στη Washington. Η Τουρκία ε, ασχολείται με τα θέματα αυτά, συζητάει τα θέματα αυτά, συζήτησε και το θέμα του Αφγανιστάν. Είναι εξαιρετικά στρατηγικό, σημαντικό εταίρος η Τουρκία για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για το Ιράν και τα πυρηνικά και για τη Μέση Ανατολή και για τον Νότιο Κάφκασο και για το Αφγανιστάν. Πολύ σημαντικός εταίρος. Προσπαθούμε να φέρουμε σε παράλληλη τροχιά την εξωτερική πολιτική της Τουρκίας με αυτήν της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν γίνει βήματα τα οποία έχουν εκτιμηθεί δεόντως από όλους τους υπουργούς εξωτερικών. Τι έχω ξεχάσει τώρα μέσα σε όλα αυτά. Αφγανιστάν και Κωσυφοπέδιο επίσης. Για το Κωσυφοπέδιο. Είναι περίπλοκο το θέμα αυτό γιατί η ανεξαρτησία του κοσφοπεδίου δεν έχει γίνει αντικείμενο αναγνώριση από όλε τι χώρε της Ευρωπαϊκής Ένωση. Παρ' όλα αυτά μπορέσαμε να κινηθούμε προς τα εμπρός. Προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε το θέμα αυτό με μια διαρθρωμένη αντιμετώπιση συνολικά το θέμα του κοσφοπεδίου και αυτό σημαίνει πως υπάρχει μια προοπτική και για την απελευθέρωση του καθεστώτος των θεωρήσεων και για το κοσυφοπέδιο. Αναγνωρίζουμε επίσης τα προβλήματα που μπορεί να υπάρχουν στη χώρα αυτή. Τώρα για το Αφγανιστάν. Εδώ ζητήθηκε η προσωπική μου άποψη για τις προσπάθειες τις οποίες κάνουμε σε πολιτικό επίπεδο στο Αφγανιστάν, όχι σε στρατιωτικό επίπεδο. Έχει κυκλοφορήσει ένα εσωτερικό έγγραφο στο Συμβούλιο γύρω από το θέμα αυτό. Το έχω συζητήσει με πάρα πολύ κόσμο για το πώς αυτή η διαθρωμένη αντιμετώπιση του Αφγανιστάν. Απαιτείται να υπάρχει μια ενιοποιημένη κοινοτική παρουσία στο Αφγανιστάν, δηλαδή κάποιος να, να παρουσιάζει και να εκπροσωπεί την Ευρωπαϊκή Ένωση στο Αφγανιστάν. Αυτό το συζητήσαμε και με την Κάθριν Άστον. Αυτά είναι τα μέσα τα οποία πρέπει να έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση εκεί. Απαιτείται όμως και καλύτερο συντονισμός μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην παρουσία του στο Αφγανιστάν. Ένα από τα θέματα που μερικές φορές κινδύνευσε να με εκνευρίσει ήταν η προσπάθεια για να καταλήξουμε στο λεγόμενο, στη λεγόμενη ε, κιανή ή μπλε βίβλο για το Αφγανιστάν. Δηλαδή ήταν πάρα πολύ δύσκολο όλες οι χώρες να βάλουν σε ένα έγγραφο το τι κάνουν στο Αφγανιστάν. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο να συγκεντρώσουμε όλες αυτές τις πληροφορίες. Δεν υπήρχαν στοιχεία, δεν υπήρχαν πληροφορίες, δεν ξέραμε τι κάνανε η Ένωση συλλογικά, συνολικά μάλλον τι έκανε στο Αφγανιστάν, αν δεν είχαμε τα στοιχεία το τι έκανε η κάθε χώρα ξεχωριστά. Και σε κάποιες συναντήσεις αναγκάστηκα να χρησιμοποιήσω πάρα πολύ σκληρή και απότομη γλώσσα. Ξοδεύουμε εκατομμύρια εκατομμυρίων σαν Ευρωπαϊκή Ένωση στο Αφγανιστάν, ασυντόνιστα ουσιαστικά. Θα πρέπει λοιπόν οι κοινοτικέ δομές να λειτουργήσουν στο Αφγανιστάν, δομές της Ευρωπαϊκής Ένωσης εννοώ και να υπάρχει ένας μηχανισμός σωστού συντονισμού της παρέμβασης έτσι ώστε σε συνεργασία με τον συντονιστικό μηχανισμό των Ηνωμένων Αθνών και με τον συντονιστικό μηχανισμό των Ηνωμένων Πολιτειών να ξέρουμε τι ακριβώς κάνουμε στο Αφγανιστάν. θα πρέπει η παρουσία μας να βελτιωθεί και στον τομέα της οικονομίας και στον τομέα της στήριξης της τάξης και αστυνόμευσης. Εγώ δεν θέλω να υπάρξει στρατιωτικοποίηση συνολικά της παρέμβασής μας εκεί και δεν θέλω τα πάντα να αναλυφθούν από τον ΝΑΤΟ. Προφανώς οι στρατιωτικές μηχανές έχουν πόρους, έχουν επίσης ε, και αρκετά μεγάλη αποτελεσματικότητα. Αλλά αυτό που χρειάζεται πρέπει να υπάρξει καλύτερος συντονισμός, μια ενιαία πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και δεν θα πρέπει να αφήσουμε τις στρατιωτικές δομές να καλύψουν όλες αυτές τις ανάγκες, γιατί βλέπουμε ότι αυτό στο τέλος δεν είναι απόλυτα ικανοποιητικό. Αυτό που αναζητούμε εδώ είναι να υπάρξει μια αποκατάσταση των κρατικών δομών της χώρας αυτής και μπορούμε να το πετύχουμε και μέσω της παρουσίας μας της πολιτικής. Και υπάρχει φυσικά και το θέμα των εκλογών. Όπως λέει η έκθεση της ομάδας που παρακολούθησε τις εκλογές εκεί, υπήρξαν σημαντικές ελλείψεις. Ε, φυσικά αυτό δεν μας εκπλήσει, είναι από τις πιο σωστές και καλύτερες εκλογικές διαδικασίες που ολοκληρώθηκαν στην περιοχή αυτή, Τατζικιστάν, Ιράν, και κάποιες άλλες χώρες οι οποίες δεν ταυτίζονται ακριβώς για να το πω έτσι απλά με την έννοια των δίκαιων εκλογών. Παρόλα αυτά και το είπα αυτό στην αρχή και το είπα και στον κύριο Καρζάη ότι δεν θα επιβιώσετε με τέτοιου είδους εκλογές. Η αξιοπιστία αυτής της εκλογικής διαδικασίας στο μέλλον δεν θα σε επιτρέψει να επιβιώσετε αν δεν βελτιωθούν τα πράγματα. Θα πρέπει λοιπόν το εκλογικό σύστημα να βελτιωθεί όσο γίνεται, εν πάση περιπτώσει να βελτιωθεί, ε, πριν από τις επερχόμενες κοινοβουλευτικές εκλογές οι οποίες προβλέπονται για τα τέλη του 2010. Απαιτούνται λοιπόν αλλαγές και θα πρέπει να βοηθήσουμε προς την ε, περίπτωση αυτή. Δεν ξέρω αν υπάρξει μια κάποια καθυστέρηση για τις κοινοβουλευτικές εκλογές. Δεν θα το αποφασίσουμε εμείς αυτό, δεν θα το αποφασίσει ούτε καν ο κύριος Καρσάη, θα το αποφασίσουν οι βουλευτές της χώρας αυτής. Και γι' αυτό σε αυτή την περίπτωση, σε αυτό το επίπεδο, ο κοινοβουλευτικό διάλογο έχει μεγάλη σημασία. Βέβαια, όταν μιλάμε για το Αφγανιστάν, μιλάμε μόνο για τον πρόεδρο Καζάη. Παντού τον πρόεδρο Καζάη ακούμε και παντού τον πρόεδρο Καζάη βλέπουμε. Αλλά παρόλα αυτά έχει και η Βουλή του Αφγανιστάν αρμοδιότητε, και δεν πρέπει να το αγνοούμε αυτό. Και ίσω ο διάλογο σε κοινοβουλευτικό επίπεδο με την Βουλή του Αφγανιστάν να είναι ένα βήμα επιπλέον που θα βοηθήσει την προσπάθεια σταθεροποίηση τη χώρα αυτή. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Περνάμε τώρα στον δεύτερο γύρο και τελευταίο γύρο των παρεμβάσεων. Ενάμιση λεπτό κύριος Μαυρονικόρας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ρωτήσω σε σχέση με, το, με τις εξελίξεις όπως αναφέρονται για την Τουρκία κατά πόσον υπάρχει μια βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση ούτως ώστε η Τουρκία να υποβάλει πραγματικές προτάσεις για τη λύση με τις γειτονικέ χώρες. Θα ήθελα να ρωτήσω κατά πόσο παρακολουθούνται οι συνομιλίες, πώς μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να βοηθήσει στις συνομιλίες και πολύ περισσότερον αν με τη δημιουργία μιας κοινή εξωτερικής πολιτικής με την κυρία Νάστον υπάρχουν οι δυνατότητες περισσότερης συμβολής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις συνομιλίες. Δεύτερο ερώτημα είναι υπάρχει τελικά μια ημερομηνία αξιολόγησης για την Τουρκία ούτως ώστε να εφαρμόσει το πρωτόκολλο της Άγκυρας μετά που έχουμε ξεπεράσει τον Δεκέμβρη. Υπάρχει ένα άλλο οριακό σημείο. Δεν ήθελα να έρθω σε σύγκρουση με τον κύριο Υπουργό, αλλά οφείλω να πω ότι μια αναφορά του με έχει βρει εντελώ αντίθετο. Η Τουρκία, η Κύπρος, η Κύπρος, η η Τουρκία γεωγραφικά ανήκουν στην Ευρώπη. Η Κύπρος είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα έλεγα για να είστε εσείς εδώ και εμείς εδώ είναι διότι σε ορισμένες κοιτίδες της γεωγραφικής Ευρώπης αναπτύχθηκαν πολιτισμοί τέτοιοι που οδήγησαν στο σημερινό ευρωπαϊκό πολιτισμό καλούμε την Τουρκία να έρθει να συμμετάσχει σε αυτόν τον πολιτισμό των δικών μας δημοκρατικών ευρωπαϊκών πολιτισμών. Thank Ευχαριστώ τον κύριο Μαυρονικόλα. Ο Γιούλαντ 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ πρόεδρε κύριε Μπίλτ. Νομίζω ότι ως ειδική Προεδρία ήταν εξαιρετική, εξαιρετικό το έργο σας. Και αν υπήρχε κάτι αντίστοιχο με τη Eurovision για τις ευρωπαϊκές προεδρίες, εγώ θα σας έδινα 12 βαθμούς, πραγματικά 12 πόντους. Νομίζω ότι η στρατηγική σας, το στρατηγικό σας όραμα για τη διέρευνα, για τη διεύρυνση, είναι πολύ υγιές και πολύ επιτυχές. Επίσης, να συγχαρώ την Προεδρία σας που αποδέχτηκε την στρατηγική για την Βαλτική. Να σας ρωτήσω για την Κούβα και για την ενδεχόμενη απελευθέρωση των σχέσεων μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Κούβας που προκάλεσε ανάμεικτα συναισθήματα όπως οι σχέσεις μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Λευκορωσίας. Ποια είναι η δική σας θέση, Υπουργέ, για τις ενδεχόμενες εξελίξεις στις σχέσεις μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Κούβας. Ευχαριστώ και τώρα ο λόγος. Thank you very much, Κυρία Άουτεν, ευχαριστώ Πρόεδρε. Είναι η Παγκόσμια ημέρα ανθρωπίνων δικαιωμάτων σήμερα και θα ήθελα να συγχαρώ την Σουηδική Προεδρία για όλες τις σχετικές προσπάθειες που έκανες και επειδή και εγώ συμμετέχω στην Υποεπιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ήταν πραγματικά εξαιρετική η συνεργασία και οφείλω να το τονίσω αυτό. Θα ήθελα να σας ρωτήσω όμως το εξής. Πώς στην καινούργια Υπηρεσία Εξωτερικών Υποθέσεων θα ενταχθούν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Δεν έχουμε επί του παρόντος σχετικές πληροφορίες για το ποιος θα προταθεί, ποιος θα διοριστεί ως εκπρόσωπος της κυρίας Άστον για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Πώς θα τονίσουμε το θέμα αυτό. Αυτό λοιπόν το θέμα της ένταξης των ανθρώπινων δικαιωμάτων είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πώς θα αποφύγουμε καταστάσεις στις οποίες έμεσα νομίζω αναφερθήκατε. Είδαμε τον κύριο Μπερλουσκόνη να πηγαίνει στην Λευκορωσία χωρίς να δίνει καμία σημασία στην αντιπολίτευση. Αυτό ακριβώς είναι τα στοιχεία που θέλουμε να αποφύγουμε. Και τρίτη ερώτηση για τη Γεωργία. Ξέρω ότι έχετε συμμετάσχει έντονα στην διαδικασία αυτή. Πώς μπορείτε λοιπόν να αναλύσετε στην παρούσα φάση της εξελίξεις τις ε, ρωσικές ε, δραστηριότητες στα κατεχόμενα ουσιαστικά εδάφη της Γεωργίας. όπου δεν υπάρχει, για παράδειγμα, πρόσβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και τώρα το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο εξετάζει τις ε, συνέπειες, όπως και το Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Πώς εκτιμάτε εσείς την κατάσταση, ευχαριστώ. Ο, ο κύριος Αγκουράκης, μισή λεπτό. Ε, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, θα ήθελα να σημειώσω τα εξή. Πρώτα απ' όλα ο κύριος Υπουργός μας μίλησε για επικείμενες συνομιλίες με τη Μολδαβία. Στη Μολδαβία όμως υπάρχει μια πολύ ασταθή πολιτική κατάσταση, όπως αγνωρίζει άριστα, ε, και γι' αυτό η συμβουλή μου είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση να μην προβεί σε καμία διαδικασία τώρα, γιατί αλλιώς, ε, κατά τη γνώμη μου, θα είναι μια ε, επέμβαση εσωτερικά της χώρας. Δεύτερο ζήτημα. Υπάρχουν τα συμπεράσματα για την συνεργασία ε, με τη Λατινική Αμερική, τη Ευρωπαϊκή Ένωση με τη Λατινική Αμερική. Ο κύριο Υπουργό δεν αναφέρθηκε ιδιαίτερα στο θέμα αυτό. Εγώ θα ήθελα ε, δύο σημεία να σημειώσω. Πρώτον, έχουμε την Αμερικάνικη παρουσία στην Κολομβία και έχει δημιουργηθεί μια ολόκληρη κατάσταση και θα ήθελα ένα σχολιασμό. Δεύτερο, έχουμε καταγγελίε για ευρωπαϊκέ πολυεθνικέ εταιρείε οι οποίε αξιοποιούν τι σχέσει με τη Λατινική Αμερική για να προβαίνουν σε απαράδεκτε καταστάσει ε, στη Λατινική Αμερική. Και τρίτον, νομίζω έχει έρθει η στιγμή να αρθεί το, η κοινή θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την Κούβα. Και τέλος, ε, νομίζουμε ότι πρέπει να παρέμβει η Ευρωπαϊκή Ένωση στις τουρκικές αρχές, διότι με ανησυχία πληροφορηθήκαμε ότι στη χώρα αυτή ετοιμάζεται η θέση ξανά εκ ε, νόμου του Κουρδικού Κόμματος, του ΔΤΠ και δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη της ε, Κομισιόν για το ζήτημα αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ τον κύριο Αγκουράκη. μισή λεπτό Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Μπίλτ. Θα ήθελα να ρωτήσω τέσσερα πράγματα σε ό,τι αφορά τη Μέση Ανατολή. Γιατί το Συμβούλιο επέλεξε να δηλώσει τις τοποθετήσεις του για τα δύο από τα τέσσερα βασικά θέματα, για τις, ε, τους επικισμούς και την Ιερουσαλήμ. Γιατί δεν ε, τοποθετήθηκε σε ό,τι αφορά τις πρόσφυγες και τις ε, διατάξεις ασφαλείας. Το Συμβούλιο δεν ε, τονίζει κάποια θέματα αποφεύγοντας κάποια άλλα. Αυτό δεν ε, είναι προς όφελος των Παλαιστινίων. Και η δήλωση του Συμβουλίου δεν δείχνει στην Παλαιστίνη ότι μπορεί να κερδίσει πιο πολλά χωρίς να δώσει και τα αντίστοιχα ανταλλάγματα προς το Ισραήλ. Αυτό δεν ε, εμποδίζει το στόχο του, του Συμβουλίου να ξεκινήσουν οι πραγματεύσεις και με τις δύο πλευρές. Γιατί δεν έγινε αναφορά στη Χαμάς και τις συνεχιζόμενες προσπάθειές της να ε, εμποδίσει την ειρηνευτική διαδικασία. Γιατί δεν ε, δηλώθηκαν αυτές οι δραστηριότητες της Χαμάς στη δήλωση του Συμβουλίου. Γιατί δεν αναφέρθηκε η κατάχρηση των ανθρωπινων, η παραβίαση των ανθρωπινών δικαιωμάτων της Χαμάς στην Γάζα. Και τέλος, γιατί το Συμβούλιο γενικά και η Συνδική Προεδρία ειδικά δεν προώθησαν μια πιο αυστηρή θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για κυρώσεις προς το Ιράν δεν έχουμε αρκετού δείκτες, δεν έχουμε αρκετέ ενδείξει ανησυχητικέ που θα δικαιολογούσαν μια πιο αυστηρή στάση για την πυρηνικό πρόγραμμα σε ό,τι αφορά και τη στάση του Ιράν για την ανθρώπινα δικαιώματα. Ευχαριστώ. Ο συνάδελφο του Λόπες, 1,5 λεπτό. Ε, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Επιτρέψτε μου να ευχαριστήσω και εγώ τον κύριο Πίλτ για τη δουλειά που έκανε κατά τη διάρκεια της Προεδρίας. Ε, και να εκφράσω και ε, την λύπη μου που δεν πετύχατε πάντα τα, αποτελέσματα που θέλατε. Θα ήθελα να ρωτήσω κάτι σχετικά με τη Λιβύη και τις ε, συμφωνίες για τη μετανάστευση. Είχατε συνομιλίες και με την Τινησία. Τι έχει γίνει ο κύριος Μπιουτικόφερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ Πίλτ, έχω τρεις ερωτήσεις. Αφγανιστάν, ε, Κολομβία και Μέση Ανατολή. Ε, Αφγανιστάν είπατε ότι η Ευρώπη θα πρέπει να μιλάει με μία φωνή και όχι να τραγουδάει σαν χοροδία. Εγώ θα ήθελα χοροδία, θα ήθελα, μία, θα ήθελα ένα ισχυρό αστυνομικό σώμα στο Αφγανιστάν εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορούσε να προσφέρει αυτή την αστυνομική εκπαίδευση που ε, ε, υπόσχεται τόσα χρόνια. Αυτό θα ήταν καλό. Θα ήθελα να ρωτήσω τι έχει κάνει η Προεδρία σας για να το αλλάξει αυτό και θα ήθελα να ρωτήσω και πόσες ακόμα Προεδρίες θα χρειαστούν μέχρι να αλλάξει αυτό ή μήπω θα έχουμε αποσυρθεί μέχρι να αλλάξει κάτι. Κολομβία. Όλο και περισσότεροι ε, συνδικαλιστές σκοτώνονται κάθε μέρα από τις οποιαδήποτε άλλη χώρα. οι Ηνωμένε Πολιτείε και ο Καναδάς ε, έχουν ε, αντιδράσει εμείς, ε, γιατί δεν το κάνουμε. Και Μέση Ανατολή την Τρίτη παρουσιάσατε τη θέση σας. Ποια είναι η στρατηγική όμως είναι η ερώτησή μου, διότι η θέση αυτή έχει προκαλέσει αντίσταση και στο Ισραήλ και στι Ηνωμένε Πολιτείε. Ε, είχατε επαφές ε, με ανθρώπους του Κογκρέσου πριν κάποιες ε, μέρες. Από την θέση αυτή πώς θα μπορέσει να δημιουργηθεί πολιτική. Ευχαριστώ κύριε Μπιουτικόφερ. Ο κύριος Σούλτς για ένα μισή λεπτό παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, ε, δικαίως ε, κοιτάτε πίσω και βλέπετε μια επιτυχημένη ε, Προεδρία. Δύο ερωτήσεις όμως σημαντικό σημείο για την Προεδρία ήταν η βελτίωση των σχέσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ρωσίας. Ε, τον έκτο κύκλο διαπραγματεύσεων είδαμε στη Στοχόλμη. Τι έχει επιτευχθεί όμως. Ε, η Ρωσία ακόμα δεν συμμετέχει στον ΠΟΕ, ο χάρτης για την ενέργεια δεν έχει επικυρωθεί. Και αν ε, μια συμφωνία εξυγχρονισμού ε, θα πρέπει να δημιουργήσει κάτι καινούριο, ε, πού βρισκόμαστε. Δεν μιλάμε πια για εταιρική, δεν μιλάμε για εταιρική σχέση. Και όσον αφορά τη Λευκορωσία, ε, θα ήθελα να ρωτήσω την ε, συμφωνία σε σχέσης ή καλής γειτονίας θα πρέπει να τη θέσουμε σε ισχύ. Τι ακριβώς γίνεται αυτή τη στιγμή. Ευχαριστώ κύριε Σούλτς. Όπως και οι συνάδελφοι θα ήθελα να σας συγχαρώ για την προσπάθεια την οποία κάνετε. Η θέση του Συμβουλίου την προηγούμενη Τρίτη για το Παλαιστινιακό ξεκαθαρίζει την ανάγκη που υπάρχει για την έβρεση μια συμφωνίας ανάμεσα στα δύο εμπλεκόμενα μέρη για την δημιουργία ενός Παλαιστινιακού κράτους, του οποίου η πρωτεύουσα θα είναι η Ανατολική Ιερουσαλήμ. Μόνιμο αίτημα, πάγιο αίτημα των Παλαιστινίων. Βέβαια θυμίζω ότι οκτώ ευρωβουλευτές της αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, με την κοινοβουλευτική ε, αντιπροσωπεία της, ε, της Παλαιστίνης δεν τους να πάνε στη Γάζα. και η ακύρωση ε, έγινε λίγες ε, ώρες μετά από την επιβεβαίωση της θέσης του ε, Συμβουλίου για τη δημιουργία ενός ανεξάρτητου Παλαιστινιακού κράτους στα σύνορα του 67. αυτή η απόφαση πραγματικά δυσκολεύει τις σχέσεις ανάμεσα στο Κοινοβουλευτικό Συμβούλιο της, των Παλαιστινίων και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γιατί ασχολούμεθα μόνο με την ασφάλεια των Ισραηλινών ενώ ε, φέτος τον χειμώνα αυτοί οι οποίοι υπέστησαν μία επίθεση και σφαγή από πλευράς των Ισραηλινών είναι οι Παλαιστίνοι. Αυτά τα δύο επίπεδα ενδιαφέροντος, οι δύο ταχύτητες αντιμετώπισης του προβλήματος είναι μία επιπλέον πηγή προβλημάτων. Συγγνώμη, ξεπεράσατε το χρόνο σας, λέει ο Πρόεδρος. Κανένας από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα δεν πήρε το λόγο γιατί βρίσκονται όλοι στην Βόνη, στην διάσκεψη της Βόνης. Ε, δύο ερωτήσεις λοιπόν θα θέσω εγώ. Η πρώτη, η θέση του Συμβουλίου για την Μέση Ανατολή. Ιδιαίτερα για το θέμα της πρωτεύουσα, το θέμα της Ιερουσαλήμ. Αυτό κατά κάποιο τρόπο προκαθόρισε το πλαίσιο μιας διαδικασίας διαπραγμάτευσης που δεν έχει ξεκινήσει ακόμα. Είναι ένα διαπραγματευτικό όπλο το οποίο έχει αρχίσει να χρησιμοποιείται. Τώρα δεύτερον, η εξωτερική υπηρεσία, το λεγόμενο διπλωματικό σώμα του πολιτικού κλάδου θα έλεγα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εμείς σαν Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θέλουμε και απαιτούμε θα έλεγα να υπάρχει δημοκρατικός έλεγχος για τον διορισμό του προσωπικού αυτής της υπηρεσίας. Η Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων και το Κοινοβούλιο μέσω αυτής έχει το δικαίωμα, θα έλεγα, συζήτησης και συναπόφασης για το καθεστώς των υπαλλήλων και εμείς σαν Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων θα θέλαμε να παρέμβουμε και εμείς στην διαδικασία επιλογής των προσώπων. Πώς ακριβώς πιστεύετε ότι μπορεί να γίνει μια τέτοια διαδικασία. Ευχαριστώ. Να, ξεκινήσω το τέλος, Πρόεδρε. Για την Κάτριν ε, Άστον που έχουμε συζητήσει το θέμα αυτό και πρέπει να σας πω ότι συμμετοποιεί απόλυτα τις ανάγκες να συνεχίσουν ε, οι συζητήσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τις ιστορικές δράσεις. Το πώς θα γίνει αυτό θα το αποφασίσει αυτή και είμαι βέβαιος ότι θα καταφέρει, ότι θα είναι σε θέση στην ακρόασή της να σας αναφέρει πολύ πιο πολλά. Τη δεύτερη εβδομάδα του Ιανουαρίου να σας πω ότι ξέρω ότι έχει αφιερώσει πολύ προσοχή σε αυτό το κρίσιμο θέμα και ότι ο διάλογος με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποτελεί τμήμα της όλης νοτροπίας ε, την οποία ακολουθεί. Θα ήταν, πιστεύω, όμω, εσφαλμένο να μπω εγώ σε λεπτομέρειες, γιατί αυτό θα πρέπει να είναι δική της αρμοδιότητα. Και θα ήθελα να πω επίσης, και αυτό είναι πολύ σημαντικό για μένα τώρα, ότι η συνθήκη της Λισαβόνας πλέον έχει εφαρμοστεί. Μέχρι 31 ε, Δεκεμβρίου θα είμαι πάρα πολύ, ε, θα επιμείνω πάρα πολύ να εφαρμοστεί η συνθήκη της Λισαβόνα σε όλες τις πτυχές, χωρίς ε, παραθυράκια. Θα πρέπει να εφαρμοστεί η συνθήκη της Λισαβόνα. Υπάρχουν κάποια θέματα, κάποια θέματα τα οποία δεν έχουν ε, επαρκώς τονιστεί σε ό,τι αφορά τη συνθήκη και γίνονται κάποιες συζητήσεις και τι συμβαίνει σήμερα και θα συμβεί και αύριο. Κάποιες φορές έχω την αίσθηση ότι περιμένετε από μένα να είμαι πρόεδρο του Συνδικάτου των Υπουργών Εξωτερικών. Ε, δεν είμαι και τέτοια πράγματα. Γιατί όλε οι προηγούμενε συνθήκε αφορούν του αρχήγου κρατών και κυβερνήσεων και του υπουργού εξωτερικών. Η συνθήκη τη Λισαβόνα αφαιρεί από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο των Υπουργών των Εξωτερικών και μιλάει για αρχηγού κρατών και κυβερνήσεων και μπορεί να πάρουν και άλλου υπουργού. Εγώ θεωρώ ότι αυτό είναι σωστό, αλλά να σα πω ότι δεν είμαι σε θέση να μπορώ να πω ότι αυτό ε, είναι κάτι που βρίσκει σύμφωνο, σύμφωνος όλους των Υπουργών Εξωτερικών. Για να το πω διπλωματικά. Αλλά είναι πολύ σημαντικό αυτό ως αλλαγή. Και γιατί? Γιατί το Συμβούλιο ουσιαστικά ασχολείται με πιο πολύ με εσωτερικές ε, υποθέσεις και Δεν θεωρώ ότι η σχέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με υποψήφιες χώρες αποφορά ε, εξωτερικές υποθέσεις. Άρα ουσιαστικά πρόκειται για επέκταση του πεδίου των ιστορικών υποθέσεων, ενώ οι εξωτερικές υποθέσεις αφορούν ουσιαστικά την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον έξω κόσμο. Άρα η λογική θα είναι ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ε, είναι και αποτελείται από τραχηγούς κυβερνήσεων και σε κάποιες περιπτώσεις θα εμπλέκει και τους υπουργού εξωτερικών, αλλά και υπουργού άλλους, ε, περιβάλλοντος για παράδειγμα. Αλλά αυτό για να σας υποδείξω που ε, έχουμε κάποιες συζητήσεις, κάποιες αμφιβολίες σε ό,τι αφορά τη συνθήκη της Λισαβόνας και άλλα θέματα τα οποία αφορούν τους ύπατους εκπροσώπους και τη σχέση τους με τους θεσμούς, τις θεσμικά όργανα σε ό,τι αφορά και το ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και εκεί έχουν τεθεί ερωτηματικά. Τώρα να απαντήσω σε ό,τι αφορά την Λατινική Αμερική, εν συντομία. Ήταν πολύ καλή σύνοδος, όπως είπατε, και με την Βραζιλία και προχωρήσαμε πολύ σε ό,τι αφορά την Ονδούρα και σε ό,τι αφορά λοιπόν ε, τη Λατινική Αμερική, Λατινική Αμερική. Είχαμε και την συνάντηση με την Κούβα. Είχαμε κάποιες ε, αναπάντηχες εξελίξεις, αλλά τελικά έλαβε χώρα αυτή η σύνοδος και είναι σαφής η γραμμή της Ένωσης ότι θέλουμε διάλογο με την Κούβα, θέλουμε σχέσεις με την Κούβα, αλλά είναι εξίσου σαφέ ότι και τα ανθρώπινα δικαιώματα αποτελούν τμήμα του διαλόγου αυτού. Δεν μπορούμε να πούμε ότι α, α συζητήσουμε, α αρχίσουμε διάλογο, αλλά να εξαιρέσουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα. Όχι, αυτό δεν είναι αποτεκτό για την Ένωση. Και αυτό αποτέλεσε ένα στοιχείο το οποίο μας ε, προκάλεσε κάποιες ε, αναταραχές μέχρι ότου έγινε αυτή η σύνοδος. Και πρέπει να σας πω ότι η Συνδική Προεδρία επέμεινε σε ότι είχε συμφωνηθεί από την Ευρώπη των 27 γιατί κάποιες χώρες ε, ε, αμφισβητούσαν τη σημασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που θα έπρεπε να έχουν τα ανθρώπινα δικαιώματα στις συζητήσεις με την Κούβα και σε ό,τι αφορά και με τις άλλες χώρες, όπως για παράδειγμα και με τη Λευκορωσία η οποία αναφέρθηκε, όπου ε, φαίνεται ότι το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων δεν είναι τόσο σημαντικό και αυτό ισχύει και σε ό,τι αφορά τον διάλογό μας με την Κολομβία που αναφέρθηκε για τον Μολδαβία. Ναι, υπάρχουν και εκεί αβεβαιότητες Πρόκειται για μια αναδυόμενη ευάλωτη δημοκρατία και υπάρχει και η σύγκρουση στην υπερδυνιστερία. Αλλά έχει σημειωθεί ένα νέο άνοιγμα για την συνεργασία με την Ένωση και νομίζω ότι ο ρόλος μας είναι να τους βοηθήσουμε. Αν δεν το πράξουμε αυτό, νομίζω ότι θα είναι πολύ λιγότερο σταθερή η κατάσταση εκεί, ό,τι και να γίνει με τις εκλογές. Γιατί η δημοκρατία πολλές φορές τίνει να είναι ασταθείς αλλά εξακολουθούμε φυσικά να τον υποστηρίζουμε πάντα είναι η κατάσταση στη γεωργία. Μία άλλη λεπτομέρεια για το θέμα της, είπα, της εκπροσώπους για τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν έχω ιδέα πρέπει να σας πω γιατί και αυτό αφορά την Κάθριν Άστον. Όλα τα θέματα εξωτερικής εκπροσώπησης θα είναι στη δική της αρμόδιότητα. Όταν λοιπόν βρεθεί, όταν αναλάβει τα καθήκοντά τη, αυτή θα τα κανονίσει για την κατάσταση στη Γεωργία. Μας ανα... ανησύχησε ιδιαίτερα η πρώτη εξεταστική επιτροπή πήγε στο Νότιο Κάφκασο και αναθεωρήσαμε την, ε, μάλλον ανανεώσαμε την εντολή τη ε, Επιτροπής ε, Παρακολούθησης εκεί και επιμείναμε σε θέματα εδαφική ακαιρεότητα. και είπαμε στον Υπουργό Εξωτερικών, όταν τον συναντήσαμε στην Νέα Υόρκη στις 27 του μηνός, το θα πρέπει να θυμάται πόσο συνεκτική ήταν πάντα η Ευρωπαϊκή Ένωση σε θέματα εδαφικής ε, ακαιρεότητας στο Βόρειο Κάφκαυσο. Όχι ότι δεν υπήρχαν προβλήματα, όπως ε, μαζικές παραβιάσεις ανθρωπινών δικαιωμάτων, αλλά όλα αυτά θα πρέπει να επιληθούν και σε ό,τι αφορά τα δικαιώματα των μειονοτήτων, σε ό,τι αφορά την εδαφική ακαιρεότητα. Και αυτό είναι εξίσου σημαντικό και στις, ε, στον Βόρειο και τον Νοτιό Όλα αυτά λοιπόν θα πρέπει να αντιμετωπιστούν από την ε, υπό το πρίσμα της λαθικής ακαιρεότητας της Ρωσίας και της Γεωργίας. Και όταν παρευρέθηκα στην Μόσχα για υπό άλλη ιδιότητα, μου δημιουργήθηκε η εντύπωση ότι είναι ανέκδοτο, κακό ανέκδοτο αυτό για τον Νότιο Κάφκασο. Επίσης, καταστήσαμε σαφές ε, προς τη Ρωσία ότι είναι σημαντικό να εφαρμόσει πλήρως τις συμφωνίες. Και αυτό περιλαμβάνει και την πλήρη απόσυρση από περιοχές όπως το Περίβη, για παράδειγμα, όπου δεν έχει ολοκληρωθεί η απόσυρση και σε ό,τι την, νότια, την Απχασία και την Νότια Οσοτία. Έχουν λειτουργήσει λοιπόν οι μηχανισμοί της Γενέβης και έχουμε καλό διάλογο με τη Ρωσία για την αποφυγή περιστατικών, οι οποίες θα μπορούσαν πολύ εύκολα να έχουν ξεφύγει από κάθε έλεγχο. Και αυτό λοιπόν θα πρέπει να το τονίσουμε ότι πέρα από τις διαφωνίες μας έχουμε καθοδρύσει πλέον ένα καλό διάλογο με τη Ρωσία. Δεν ε, αναμένω άμεση επίλυση των ζητήματων αυτών. Αναμένω ε, διαβούλευση για την αντιμετώπιση των θεμάτων αυτών μέχρι να αλλάξει κάπως η κατάσταση και να περάσουμε στην επίλυση των συγκρούσεων. Αλλά παραμένει πολύ σημαντικό το θέμα και φυσικά δεν χρειάζεται να σας πω ότι έχουμε και στενό διάλογο με τους εκπροσώπους της Γεωργίας. Χαίρομαι που αναφέρθηκε και η πολιτική για την Βαλτική. Δεν αποτελεί θέμα εξωτερικών υποθέσεων, αλλά ασφαλώς αποτελεί κληροδότημα της Σουηδικής Προεδρίας για τη Λατινική Αμερική. Ούτε αυτό αφορά ιδιαίτερα την Σουηδική Προεδρία, αλλά θα γίνει μια σύνοδο στη Μαδρίτη την Άνοιξη μεταξύ εκπροσώπου τη Λατινική Αμερική και τη Καραϊβική και τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα βλέπετε ότι στην έμφαση τη Σουηδική Προεδρία ήταν ο στρατηγικό διάλογο με αναδυόμενες δυνάμεις και νομίζω ότι τους επόμενους έξι μήνες θα δούμε έντονη εκπροσώπηση της Λατινικής Αμερικής, το οποίο θεωρώ ότι είναι θετικό και το καλωσορίζω για την ε, Ρωσία και πάλι. Εν συντομία, ήταν καλή η συνάντηση με τη Ρωσία στη Στοκχόλμη, δεν τίθεται θέμα γι' αυτό. Αλλά θέλουμε και συγκεκριμένα αποτελέσματα. Ποια είναι λοιπόν τα συγκεκριμένα αποτελέσματα. Η διαπραγμάτευση νέας συμφωνίας, η οποία προχωράει στα πλαίσια του ΠΟΕ και λάβαμε ενθαρρυντικές ε, ενδείξεις από τον πρόεδρο με σε ό,τι αφορά τον ΠΟΕ. Αλλά δεν ε, μπορώ να παραλείψω να πω ότι ο Πρωθυπουργό Πούτιν εμφανίστηκε πριν από δύο εβδομάδες ε, στην τηλεόραση και η διατύπωσή του ήταν διαφορετική. Ο πρόεδρος Μετβέντεφ μίλησε για προσχώρηση στον ΠΟΕ το συντομότερο δυνατόν, ενώ ο Πρωθυπουργό Πούτιν το ανέφερε αυτό ως μακροπρόθεσμο σχέδιο. Δεν ξέρουμε όμως τι θα γίνει. Απλά επαναλαμβάνουμε ότι θα θέλαμε να τους καλωσορίσουμε το συντομότερο δυνατόν στον ΠΟΕ και ότι θέλουμε πιο βαθύ διάλογο σε ό,τι αφορά θέματα ενέργειας αλλά και σε όλα τα άλλα θέματα και έχουμε συμφέρον να εξυγχρονιστεί η Ρωσία και να αναπτυχθεί το κράτος δικαίου. Και ο Μετβέντεφ δεσμεύτηκε στο κράτος δικαίου, αλλά φυσικά υπάρχουν και κάποια θέματα εφαρμογής τα οποία δεν είναι ασήμαντα και αυτά και θα πρέπει να αντιμετωπιστούν. Αλλά η προώθηση του διαλόγου θα έχει ως αποτέλεσμα θετικά αποτελέσματα για τη Λιβύη. Να ομολογήσω ότι δεν παρακολουθώ όλα τα θέματα, αλλά θα γίνει στις 17 Δεκεμβρίου ε, επόμενο γύρο διαπραγματεύσεων και θα τεθεί και το θέμα της μετανάστευσης στην ατζέντα. Και από ό,τι μου είπαν, οι διαπραγματεύσει αυτέ είναι δύσκολε και δεν μου προκαλεί καθόλου έκπληξη το γεγονό αυτό. Μη μου ρωτήσετε τίποτα άλλο, γιατί δεν ξέρω και τίποτα άλλο να σα πω για το θέμα αυτό. Ύστερα, για το Αφγανιστάν και για την αστυνομία, την αστυνομική δύναμη. Συμφωνώ ότι καταφέραμε να αυξήσουμε την, την αστυνομική μας δύναμη. Έχω αποστείλει επιστολές, έχω μιλήσει με τους υπουργούς και αυτό μας οδήγησε στο αποτέλεσμα να έχουμε αυξήσει τις αστυνομικές μας δυνάμεις. τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τις δεσμεύσεις μας δεν έχουμε ακόμα αποστείλει δυνάμεις. Θα πρέπει να το συζητήσω και με την Κάθριν Άστον για να συνεχίσει τις προσπάθειες αυτές στον κλάδο αυτό για να αυξηθεί η αστυνομική η δύναμη. Τώρα, αν θα το πετύχουμε αυτό, θα το δούμε. Θα πρέπει να εκπληρώσουμε τις δεσμεύσεις μας για τις κυρώσεις στο Ιράν. Απάντησα. Δεν έχουμε φτάσει στο σημείο αυτό. Και βρισκόμαστε σε στενό διάλογο με τους Αμερικανούς ομολόγους. Θα πρέπει να ακολουθήσουν και άλλες διαβουλεύσεις και θα συμπεριληφθεί το θέμα αυτό, φαντάζομαι, στο επόμενο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων και έχουμε κάνει σημαντικές αναλύσεις για να εξετάσουμε και τις δυνατότητες και τα προβλήματα με τα οποία βρισκόμαστε αντιμέτωποι. Να πω ότι έχω κάποιες εμπειρίες ό,τι αφορά πολιτική κυριώσεων σε διάφορους τομείς και είναι ένας τομέας τον οποίο εύκολα μπορούμε να συζητήσουμε, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο στην εφαρμογή. Θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί στην εφαρμογή, γιατί είναι πολύ δελεαστικό να αυτό αυτοπυροβοληθούμε αν θέλετε, αλλά θα πρέπει ασφαλώς να το αποφύγουμε αυτό. Δεν λέω ότι είναι και αδύνατον, αλλά να ξέρει κανείς ακριβώς τι κάνει, να ξέρει ποιον στόχο επιδιώκει. Ιδάλλως κινδυνεύουμε να είμαστε αντιπαραγωγικοί ή να καταστούμε απλά, αν θέλετε, γραφικοί, να, είμαστε, να παραμείνουμε απλά σε ρητορικό επίπεδο. Θα πρέπει λοιπόν να επιτύξουμε εξαιρετική επιφύλαξη και προσοχή χρησιμοποιώντας όλη την ευφύεια μας για τη Μέση Ανατολή και πάλι. Και τέλος, πολλά θέματα παραμένουν ανοιχτά και θα πρέπει να αντιμετωπιστούν. Το θέμα των προσφύγων, το θέμα της ασφάλειας των συνόρων, της Ιερουσαλήμ, όπως σας είπα, ασχοληθήκαμε πάρα πολύ ασχοληθήκαμε πάρα πολύ με το θέμα των προσφύγων και σε θέματα ασφαλείας τα οποία θεωρούμε σημαντικά, όπως και οι Αμερικανοί. Έχουν ξεκινήσει λοιπόν οι εργασίες προς αυτή την κατεύθυνση και στο επίκεντρο είναι το θέμα των επικισμών και των συνόρων, γιατί αυτά είναι θεμελιώδη ζητήματα. Αν επιτύχουμε συμφωνία για τα σύνορα, για παράδειγμα, βάσει τη συμφωνία του 67, συμπεριλαμβανομένη τη Ιερουσαλήμ, έχουμε επιλύσει πάρα πολλά είδη και τα υπόλοιπα, αν θέλετε, θα τρομολογηθούν. Και γι' αυτό είναι σημαντικό να εκφραστούμε ως προς αυτή την κατεύθυνση. Μου είπατε ότι ωραία, καλή η πολιτική, αλλά που είναι η στρατηγική. Καλή ερώτηση. Γιατί με πάσα ειλικρινία σας είπα ότι υφίσταται η Ευρωπαϊκή Ένωση και είμαστε παρόντες, αλλά ο μηχανισμός μας ε, είναι καλύτερος στην έκδοση αποφάσεων παρά στην ε, έκδοση συγκεκριμένης στρατηγικής, αλλά βελτιωνόμαστε και προς αυτή την κατεύθυνση. Να βρούμε λοιπόν κάποιες παραμέτρους και να υποδείξουμε το, την κατεύθυνση την οποία ακολουθούμε. Αυτό είναι σημαντικό, γιατί από τη στιγμή που θα οριστούν οι παράμετροι, από τη στιγμή που θα οριστούν οι στόχοι και θα ενθαρρυνθεί ο διάλογος, έχουμε κάνει ένα σημαντικό βήμα. Έχουμε συνεργαστεί πάρα πολύ στενά με τους Αμερικανούς. Κάποιοι στο Κογκρέσιο διαφωνούν. Ναι, προφανώς είναι αμφιλεγόμενο το θέμα και προφανώς και εδώ, μετά από αυτά που άκουσα, δεν μπορώ να πω ότι είναι ε, ομόφωνη η άποψή σα για τη Μέση Ανατολή. Έτσι έχουν τα πράγματα, αλλά παρόλα αυτά θα πρέπει να αναπτύξουμε μια στρατηγική, μια πολιτική για να οριστούν από ευρωπαϊκής πλευράς κάποιες παράμετροι και το γεγονός ότι βρέθηκαν αυτές οι παράμετροι είναι φετικό για την έναξη των διαπραγματεύσεων να είμαστε σαφείς ε, για το θέμα της Γάζας, να υποστηρίξουμε τους Παλαιστινίους. Και ξέρουμε ότι το θέμα της Γάζας συνδέεται και με άλλα θέματα. Και μετά να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις. Νομίζω ότι θα πρέπει να διαδραματίσουμε ένα ρόλο στις διαπραγματεύσεις αυτές. Αλλά τον πρώτο ρόλο προφανώς θα παίξουν οι ΙΠΑ. Δεν έχουμε φτάσει όμως στο σημείο αυτό ακόμη. Δεν έχουν ξεκινήσει τέτοιες συνομιλίες. Αλλά νομίζω ότι η δήλωσή μας, η πρόσφατη δήλωσή μας ήταν επισημαντική για την Ιερουσαλήμ. Προφανώς αποτελεί αυτό θεμελιώδες σύντημα. και είναι και δύσκολο θέμα αυτό γιατί έχουμε, αν θέλετε, τα συναισθήματα των τριών μεγάλων δογμάτων, αβραμικών δογμάτων ε, του κόσμου και χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή για αντιμετώπιση του θέματος αυτού. Γιατί είναι έντονα τα συναισθήματα μεταξύ μουσουλμάνων, χριστιανών και Εβραίων σε όλο τον κόσμο. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει η πόλη αυτή να είναι μια πόλη για όλους και αν διαμορφωθούν δύο κράτη, το οποίο και ελπίζουμε, αυτή η Ιερουσαλήμ θα πρέπει να είναι η πρωτεύουσα και των δύο κρατών. Και θα πρέπει φυσικά τα δύο μέρη να λύσουν τις υπόλοιπες λεπτομέρειες μεταξύ τους. Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ. Η συνάντηση ήταν νομίζω καρποφόρα, ενδιαφέρουσα. Υπήρξαν πάρα πολλές ερωτήσεις και αρκετές από αυτές ήταν δύσκολες και δείξατε ακριβώς την δυνατότητά σας να δίνετε τις πληροφορίες ε, εκεί που πρέπει. Ίσως κάποιοι να έχουν μείνει με ορισμένα ερωτηματικά, αλλά η πολιτική και ιδιαίτερα η εξωτερική πολιτική είναι σε μόνιμη εξέλιξη, αλλάζει συνεχώς και θα υπάρξουν πράγματι και περισσότερες ενέργειες από πλευράς μας και θα συνεχίσουμε το διάλογο μαζί σας μέχρι το τέλος της Προεδρίας σας. Σας ευχαριστώ ιδιαίτερα. Σε λίγα λεπτά σε αυτή την αίθουσα θα ξεκινήσει η συνεδρίαση της Υποεπιτροπής για θέματα ασφάλειας και άμυνας. Εμείς θα συνεδριάσουμε την 17η του μηνός στο Στρασβούργο. Ah,